Um, Καλησπέρα σας, συνάδελφοι. Περίμενα λίγα λεπτά, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το θέμα. Τρεις η ώρα την Δευτέρα ταξιδεύει ο κόσμος και έχουμε πολύ σημαντικά θέματα για το πακέτο ασύλου στις 3 η ώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν όσους ήρθατε. Θα ξεκινήσω συνήθως με τις ανακοινώσεις ε, και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, εγκρίνεται. Για τα γλωσσικά, δανέζικα, μαλτέζικα, κροατικά και Ιρλανδικά δεν θα έχουμε και μετά έχουμε την έγκριση των συστάσεων των συντονιστών ορισμό εισηγητών. Ο κύριος Σόγκορ του ΕΛΚΑ έχει οριστεί εισηγητής για την ενιαία ψηφιακή πύλη για παροχή πληροφοριών βοήθειας και επίλυσης προβλημάτων. Εγκρίνεται, ναι, ωραία, ευχαριστώ. Μετά πράξεις κατεφαρμογή εφαρμογή και κατεξοδότηση. 23 Νοεμβρίου το Κοινοβούλιο έλαβε το σχέδιο εφαρμοστικής απόφασης ε, για την απόφαση 2015-2403 για κοινές κατευθυντήριες γραμμές ε, για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων έτσι ώστε αυτά να καταστούν μονίμως ε, μη λειτουργικά. Η βασική οδηγία είναι η 2017-853 που τροποποιεί την οδηγία 91-477 ΕΟΚ για τα πυροβόλα όπλα. Αυτό είναι σύμφωνος με το άρθρο 54, τα έχουν λάβει όλα τα μέλη της Επιτροπής μας ε, και υπήρχε μια ιστορική προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων. Αν υπάρχει κάποια αντιρρήση, ενημερώστε την γραμματεία πριν από τις 8 Δεκεμβρίου. Και τέλος υπάρχει η ηλεκτρονική ψηφοφορία αύριο 5 και 45. Παρακαλώ να φέρετε τις κάρτες σας. Και περνάμε τώρα στο βασικό μας θέμα απόψε για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, συνάδελφοι, επ' αυτού του θέματος οι συντονιστές αποφάσισαν να γίνει μια συζήτηση για το που ακριβώς βρισκόμαστε πολιτικά στο όλο θέμα αυτό. Θέλω απλά να σας πενθυμίσω το που βρισκόμαστε και την σημασία αυτού του πακέτου. Υπάρχουν 8 εισηγητέ της Επιτροπής μας. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για ένα τεράστιο εγχείρημα. Και βεβαίως έχει και πολιτική σημασία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, αναδιατύπωση Eurodac, αναδιατύπωση Δουβλίνου, κανονισμός διαδικασιών ασύλου, το πλαίσιο μεταγκατάστασης ε, και ο κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών προέλευσης. Οπότε, ο στόχος της σημερινής ε, συζήτησης δεν είναι να μπούμε σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειε για τα κείμενα του κάθε νομοθετήματος, γιατί είναι και αδύνατον. Αυτό το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε πού πηγαίνουν διάφορα στοιχεία του πακέτου και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδελφούς της Κομισιόν και του Συμβουλίου να εστιάσουν σε αυτό να μην μπουν σε λεπτομέρειες τις οποίες ξέρουμε. Κάποιοι εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές είναι εδώ. Το ερώτημα είναι προς τα πού πηγαίνουν αυτοί οι φάκελοι πολιτικά που βρισκόμαστε λίγο πριν τα Χριστούγεννα και τι μπορούμε να περιμένουμε στα πολιτικά πολύ ευαίσθητα αυτά ζητήματα και σε τι κατάσταση βρίσκεται το πακέτο αυτό. Να υπενθυμίσω συναδέλφους ότι τον Μάιο και τον Ιούλιο η Κομισιόν έκανε 7 νομοθετικές προτάσεις σε δύο πακέτα για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου πέρα από την πρόταση για ένα κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών ε, που πρότεινε η κυρία Γκυγιόμ ήδη από το 2015 και όπου ανεστάλησαν οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο για να περιληφθεί ο κατάλογος στον κανονισμό διαδικασίων ασύλου. Έκτοτε, σε έξι από αυτά τα θέματα το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει διαπραγματευτική εντολή με πιο τελευταίο τον κανονισμό του Δουβλίνου. Και θα έρθει και η συνάδελφος αργότερα. Οπότε, οι προτάσεις ε, είναι σε διαφορετική φάση της νομοθετικής διαδικασίας. Η πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σύλλου έχει φτάσει στην φάση μιας προσωρινής συμφωνίας. Έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για την αναδιατύπωση του Eurodac ε, και τον κανονισμό περί ε, όρων. Το Συμβούλιο όμως δεν έχει συμφωνήσει σε μια διαπραγματευτική εντολή για τις συνθήκες υποδοχής, ε, τον κανονισμό διαδικασιών ασύλου και των κανονισμών διατύπωσης του Δουβλίνου. Οπότε βλέπουμε μια ανισορροπία η οποία γυρεί σοβαρά ερωτήματα για την βούληση και την ικανότητα να ολοκληρωθεί αυτό το πακέτο ασύλου. Οι προτάσεις βεβαίως είναι αλληλένδετες και ε, δεν υπάρχει απαραίτητη σύνοχη. Και αναμένουμε τις απόψεις ε, Κομισιόν και Συμβουλίου. Οπότε Τώρα δεν θα ακούσουμε όλες τις λεπτομέρειες όλων των προτάσεων. Θα ακούσουμε μια πολιτική παρουσίαση, θα έλεγα, από την Κομισιόν και το Συμβούλιο για το που βρίσκονται και μετά ελπίζω να ακούσουμε και τους συζητητές. Θα δώσω τώρα πρώτα τον λόγο στην Κομισιόν στον κύριο Ράιαν, επικεφαλής ε, της αρμοδιασμόναδας της Κομισιόν και έχετε τον λόγο για 7 λεπτά. Εντάξει, ξέρω ότι δεν ακούγεται πολύ, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις. Και θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια από αυτά τα ζητήματα. Οπότε, πείτε μας πώς έχει η στρατηγική και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πακέτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σαφή γίνεται. Θα ήθελα να σα ανακεφαλώσω το πού ακριβώ βρισκόμαστε στι διαπραγματεύσει. Μετά από τι 7 προτάσει, η Κομισιόν ανέλαβε να μεταρρυθμίσει γενικά το σύστημα των δέσμη μέτρων. Και θα αναφερθώ και στη σχέση ανάμεσα στο σχέδιο των προτάσεων, επί των οποίων συζητάμε. Πολλέ, ε, τόσο από τεχνική όσο και πολιτική σκοπιά, ε, παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Και τέλο, θα σα αναφέρω ποιε κατά την άποψή μα ε, είναι οι επιπτώσεις ε, ε, για τον χρόνο αλλά και για τις συνέπειες ε, των διαπραγματεύσεων μετά την ολοκλήρωσή τους. Ας δούμε λιγάκι τα μεμονωμένα εργαλεία που υπάρχουν. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά τα οποία είπατε εσείς. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στους, στα θέματα, στους φακέλους όπου έχουμε σημειώσει πρόοδο. Οι συνομοθέτες έχουν επιτύχει ευρεία πολιτική συμφωνία ε, για την ε, επαναφορά της εντολής προς την υπηρεσία. Αυτό έγινε τον Ιούνιο αυτού του έτους και ολοκληρώθηκαν εργασία σε τεχνικό επίπεδο ε, στις αιτιολογικές σκέψεις. Η διασύνδεση με τις άλλες προτάσεις και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί και μάλιστα στο εγγύς μέλλον. Όσον αφορά τη Eurodac, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τα δύο ενέκριναν τις εντολές που τους εδόθησαν και είχαμε το φθινόπωρο τρεις τριμερείς διαλόγους ε, τον Νοέμβρη και, είχαμε και τριμερι, έχουμε τριμερή διάλογο αυτή την εβδομάδα και την επόμενη στο Στρασβούργο. Οι προσδοκίες μας είναι ότι θα καταστεί δυνατόν να επιτύχουμε πολιτική συμφωνία και αυτό πριν από τα τέλη του έτους. Δηλαδή ε, μέχρι τέλος του 2017. Υπάρχουν βέβαια πολλά σημαντικά θέματα που πρέπει να επιληθούν συμπεριλαμβανομένης και της περίοδου αποθήκευσης των δεδομένων και ε, της διάρκειας ε, κατά την οποία θα υπάρχει πρόσβαση ε, στην ισχύ και στις νομοθετικές πράξεις. Υπάρχουν, έχουμε τους δύο οργανισμούς, τους δύο θεσμούς που έχουν τοποθετηθεί και είχαμε ήδη τρεις, ε, δύο τριμερείς διαλόγους, έναν επίσης αυτή τη βδομάδα και άλλον ένα μετά από κάποιες εβδομάδες. Ακόμα δεν έχουν συμφωνηθεί οι συμβαστικές προτάσεις, σημειώνεται όμως σταθερή πρόοδος και νομίζω ότι υπάρχει ε, σύγκληση απόψεων σε μεγάλο βαθμό ανάμεσα στους συνομοθέτες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τις προσδοκίες εναρμόνισης τόσο για τα κριτήρια της επιλεξιμότητας όσο και το περιεχόμενο της προστασίας προς τους δικαιούχους. Όσον αφορά την οδηγία περί ε, προϋποθέσεων υποδοχής, η δουλειά στο Συμβούλιο έχει προχωρήσει αρκετά καλά και αναμένουμε το Συμβούλιο να καταλήξει σε μια μερική γενική συμφωνία την Τετάρτη αυτής της εβδομάδος. Και κατόπιν πιστεύουμε ότι οι τριμερείς διάλογοι θα ξεκινήσουν μετά από κάποιες εβδομάδες. Επ' αυτού του θέματος. Για να ανακεφαλαιώσω λοιπόν, επί της ουσίας νομίζω υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σύμπτωση απόψεων ανάμεσα στους θεσμούς, αλλά υπάρχουν βέβαια και κάποια σημεία όπου υπάρχει διάσταση απόψεων, κυρίως όσον αφορά το χρόνο, χρονικό διάστημα που θα υπάρχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την κράτηση των ανηλίκων ε, και κάποια μέτρα που αφορούν στην υποδοχή για να αποφευθούν δευτερογενείς μετακινήσεις. Όσον αφορά τον κανισμό για διαδικασία διαδικασία περί ασύλου. Εδώ μικρότερη πρόοδος, ε, βραδύτερη λόγω της περιπλοκότητας του εργαλείου. Βέβαια ε, στο Συμβούλιο έχει σημειωθεί πολύ καλή δουλειά κατά τη διάρκεια της Εστονικής Προεδρίας και τώρα έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τη δεύτερη ανάγνωση ε, του κειμένου, ενός κειμένου συμβαστικού που κατέθεσε η Προεδρία. Κατά τη διάρκεια συζήτησης για το συμβαστικό κείμενο δώσαμε σημασία στις διατάξεις που αφορούν Στι στις ασφαλείς ε, τρίτες χώρες ε, μετά βέβαια από οδηγίες που λάβαμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου και προσβλέπουμε στο ότι οι διαπραγματεύσεις ε, στο Συμβούλιο θα ολοκληρωθούν τουλάχιστον κάποια στιγμή την άνοιξη του επόμενου έτους. Και όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, Χρειάζεται λίγος περισσότερος χρόνος για το Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί, αλλά αναμένεται ότι θα κατατεθεί σχέδιο έκθεσης μέχρι το τέλος του, του Και όχι μόνο να κατεθεί να εγκριθεί η έκθεση μέχρι τέλος έτους. Πάμε στη Συμφωνία του Δουβλίνου. Αυτό είναι το πιο δύσκολο θέμα από όλα. Οι συζητήσεις να το πω αλλιώ, υπήρξε μια ανάγνωση στο Συμβούλιο σε επίπεδο εργασία, τεχνικό επίπεδο και ε, τα τελευταία χρόνια είχαν λάβει η χώρα πολλές ε, διμερείς ε, συζητήσεις σε ανώτατο επίπεδο Νομίζω λοιπόν όλοι γνωρίζουν ότι εκείνο το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για ορισμένα κράτη-μέλη είναι η συμπερίληψη στην πρώτη κομισιόν της ε, υποχρεωτικής ε, επαναγκατάστασης, relocation, η περίφημη πρόταση να ε, εγκαθίστανται αλλού οι πρόσφυγες από τη στιγμή που τα έχει επιτευχθεί ένα ανώτατο όριο. Το Κοινοβούλιο δέχτηκε αυτή την εντολή και είναι σαφές πλέον ότι το χρονικό διάστημα για να υπάρξει συμφωνία σχετικά με το στοιχείο της αλληλεγγύης ε, σχετικά και με τη μεταρρύθμιση δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τόσο για το χρονικό διάστημα όσο και για το περιεχόμενο αυτής της αλλαγής. Όσον αφορά ε, το πλαίσιο της επαναγκατάστασης, της resettlement, ε, νομίζω ότι επιτεύχθηκε κοινή θέση από το Συμβούλιο. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα έγινε αυτό και το Κοινοβούλιο κατέληξε σε θέση τέλη Οκτωβρίου. Περιμένουμε ο πρώτος τριμερής διάλογος να λάβει χώρα στις 13 Δοδεκάτου. Και πάλι λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό ε, σύμπτωση απόψεων των θεσμών. Είναι, συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο και κάθε δύο χρόνια να καταρτίζεται και ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη διάσταση ε, των φιλοδοξιών που πρέπει να έχουμε αλλά και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ε, το Συμβούλιο λέει να υπάρξει εφαρμοστική πράξη και το Κοινοβούλιο λέει τα μέτρα και τα σχέδια να εγκρίνονται με κατεξουσιοδότηση πράξης. Η τελευταία πρόταση την οποία και εσείς ε, υπενεχθήκατε, κατ' ουσίαν οι διαπραγματεύσεις ανεστάλησαν ε, λόγω της ε, πρότασης της Κομισιόν για ένα κανονισμό σχετικά με τη διαδικασία περιχωρήγησης ασύλου. Αυτός ο κανονισμός θα αναλάβει και θα υιοθετήσει ό,τι ισχύει. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι, υπάρχουν προκλήσεις, είναι δύσκολα τα θέματα, έχει όμως σημειωθεί και ουσιαστική πρόοδος. Και θα ήθελα να πω τώρα κάτι σχετικά με τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα διάφορα θέματα. Σας είπα ότι υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στα θέματα και πρέπει πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω κατά την άποψη της Κομισιόν όλες οι προτάσεις πρέπει να θετηθούν έτσι ώστε να έχουμε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ο χρόνος μετράει περισσότερο και όχι το να επιλεγούν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Ε, δεν πρόκειται για επιλογή πολιτικών. Και κάτι άλλο, πρακτικής φύσεως. Ε, θέλω να πω το εξή ε, να διασφαλίσουμε και τη συνέπεια ανάμεσα στις διάφορες προτάσεις, να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρηθεί η συνέπεια στις διαπραγματεύσεις και με τους άλλους θεσμούς, γιατί υπάρχουν ε, πολλές πρακτικές δυσκολίες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελήφθησαν κάποιες αυθαίρετες αποφάσεις πριν από 15 χρόνια από τους νομοθέτες ε, να υπάρχουν διαφορετικά εργαλεία στο σύστημα χορήγησης ασύλου. Δεν είναι όμως πολύ λογικά όλα αυτά. Σας είπα ότι είναι λιγάκι αυθαίρετα και γι' αυτό εξακολουθούμε ε, ακόμα να παλεύουμε με αυτή την απόφαση πρακτικά το τι δηλαδή μπορούμε να κάνουμε υπάρχουν τακτικές ε, συναντήσει των εμπειρογνωμών που ασχολούνται με αυτό το θέμα για να μπορέσουν να διασφαλίσουν ότι θα διατηρηθεί η συνοχή και η συνέπεια. Επί τη ουσία, επιτρέψτε μου να επισημάνω ορισμένου βασικούς τομείς όπου η συνέπεια και η διασύνδεση των θεμάτων είναι πολύ σημαντική. Πρώτα απ' όλα, αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι όσον αφορά τι διατάξει για την απόφαση δευτερογενών μετακινήσεων, αυτή η απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κανονισμό του Δουβλίνου, για τους κανονισμούς ε, περί διαδικασίας ασύλου και περί υποδοχής ε, και όχι τόσο ε, μεγάλη σημασία για τα κριτήρια. Όλα αυτά προσπαθούν να συστήσουν ένα κοινό πλαίσιο να υπάρχουν σαφείς υποχρεώσεις από πλευράς ε, ετούντων να καταβάλουν, υποβάλουν την αίτησή τους ε, στην πρώτη χώρα όπου ε, φτάνουν και εκεί να παραμένουν. Να είναι επίσης σαφές όσον αφορά τις συνέπειες που προκύπτουν από τις μετακινήσεις των ετούντων άσυλο. Μετακινήσεις τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο, αυτό αφορά τόσο διαδικασία όσο και την υποδοχή τους. Επίσης, διευκρινίζονται υποχρεώσεις των κρατών μελών, ε, είναι υποχρεωμένα να αποτρέπουν δευτερογενείς μετακινήσεις. Άρα, δηλαδή, οι διαπραγματεύσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να ρυθμιστούν ταυτόχρονα σε όλα ε, τα διαφορετικά εργαλεία που υπάρχουν. Ένα άλλο παράδειγμα όπου υπάρχει σαφή διασύνδεση ανάμεσα στα εφιστάμενα εργαλεία αφορά στη μεταχείριση κυρίως των ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων ατόμων που έχουν ε, ανάγκη υποδοχής. Ε, νομίζω ότι ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράδειγμα αφορά ε, στην ε, θεσμική παρακολούθηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλα τα εργαλεία που προανέφερα. Όταν πρόκειται για την εντολή ε, του ανθρώπου που προσέχει τους ανήλικους, ε, για πόσο χρονικό διάστημα θα είναι αρμόδιος. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην εντολή προς την υπηρεσία και το νομικό πλαίσιο. Ε, εδώ μπορώ να φέρω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Τώρα η υπηρεσία έχει τη συγκεκριμένη εντολή να συστήνει, να συντάσει εκθέσεις ε, για τις χώρες προέλευσης και αυτό επηρεάζει σαφώς τον κανονισμό περί ε, χαρακτηριστικών. Qualification Regulation. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι όσον αφορά τις ασφαλείς σε τρίτες χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την υπηρεσία να συγκεντρώσει πληροφορίες που είναι σημαντικές για να μπορεί να αποφασίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον θα συμπεριλάβει αυτές τις τρίτες χώρες στους καταλόγους Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασφαλείς τρίτες χώρες. Τώρα, για το μέλλον, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι 18 μήνες μετά την υιοθέτηση των προτάσεων είμαστε σε τελείως διαφορετική θέση όσον αφορά τα διάφορα εργαλεία. Και νομίζω ότι θα χρειαστούμε όμως ακόμα κάποιο χρόνο για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, κυρίως όσον αφορά στον κανονισμό του Τουβλίνου και στον κανονισμό περί διαδικασιών χορήγησης ασύλου. Ε, το περιεχόμενο είναι πολύ ευαίσθητο και είναι και περίπλοκο. Επίσης υπάρχουν δύο εργαλεία όπου σε μεγάλο βαθμό έχουμε συμφωνήσει επί του περιεχομένου. Είμαστε κοντά στο να συμφωνήσουμε. Πρόκειται για την υπηρεσία και για τις συμφωνίες περί Eurodac. Από πλευράς Κομισιόν νομίζω ότι ήταν λάθος να μην κεφαλοποιήσουμε ε, το ότι έχουμε φτάσει τόσο κοντά σε αυτές τις ε, σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ε, επί της ουσίας, επί του περιεχομένου έχει ήδη προκύψει συμφωνία και νομίζω θα μπορούσαν να προκύψουν βραχυπρόθεσμα λειτουργικά ωφέλη.

Τώρα πλέον έχουμε ε, καλύτερη εντολή για την υπηρεσία, συγκεκριμένους πόρους που διαθέτει η υπηρεσία ε, και επίσης ε, υποστήριξη που μπορεί η υπηρεσία να προσφέρει προς τα κράτη-μέλη. Το ίδιο ισχύει και για τον κανισμό Eurodac. Νομίζω ότι ήδη μπορεί να αρχίσει να ισχύει για την αντιμετώπιση της νομότυπης μετανάστευσης για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του νόμου. Στις 27 Σεπτεμβρίου όταν εγκρίναμε ε, την Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεθάρνε τους συνομοθέτες να προχωρήσουν, να ολοκληρώσουν τη συμφωνία για αυτά τα δύο εργαλεία. Διότι πιστεύει η Επιτροπή ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία ίσως πρέπει να τροποποιηθούν, αλλά αργότερα, μετά την έγκριση της συμφωνίας, γιατί θα ήταν ντροπή εντωμεταξύ να μην αποφεληθούμε από την επίτευξη της συμφωνίας. Ευχαριστούμε πολύ και για το περιεχόμενο και τα περιστρατηγικής που ενδιαφέρουν τους συναδέρφους σίγουρα. Οι πρόσωποι του Συμβουλίου τώρα παρακαλώ. Σομπλές και Λουίσου. Σας ευχαριστώ πολύ που μας βοηθάτε. Λοιπόν και εσείς τώρα. Ίσως 7-10 λεπτά το πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, νομίζω ότι μπορώ να είμαι σύντομη, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι ανέφερε σε βάθος σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή η υπόθεση, ποια είναι τα ζητήματα που παραμένουν σε κρεμότητα, ποια έχουν ήδη ξεκαθαριστεί. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε να έρθουμε σε αυτήν εδώ τη συνεδρίαση και μας επιτρέπετε έτσι να σας παρουσιάσουμε το έργο μας και πώς να διασφαλίσουμε τη συνοχή τελικά, γιατί περί αυτού πρόκειται, ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Όπως είπε και ο υπουργό μας όταν ήρθε τον Ιούλιο εδώ στην Επιτροπή σας, ο κύριος στόχος της Προεδρίας είναι να πετύχει, να πετύχει όσο γίνεται περισσότερη πρόοδο στις διάφορες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τη μεταρρύθμιση. Χτίζοντας πάντως στο έργο των προηγούμενων προεδριών, κάτι το οποίο και κάναμε. Γι' αυτό και προχωρήσαμε τις νομοθετικές προτάσεις του πακέτου. Τέσσερις εντολές έχουν ήδη συμφωνηθεί πάντως και κατά τη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας και άλλων, ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον ελπίζουμε να μπορέσουμε να κλείσουμε και πέμπτη εντολή όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής και ελπίζουμε ήδη τώρα την Τετάρτη να το πετύχουμε αυτό. Τώρα για τη συνοχή των ε, υποθέσεων αυτών μεταξύ τους. Πράγματι έχουν γίνει προσπάθειες, η πρόκληση ήταν μεγάλη, αλλά νομίζω ότι καταφέραμε να παραμείνουμε στην ιδέα για το ότι ό,τι αποφασίσουμε θα μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη και θα υπάρχει συνέπεια μεταξύ των διαφόρων φακέλων. Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και βασιστήκαμε στη Μαλτέζικη Προεδρία, η οποία είχε ήδη εντοπίσει τα κύρια ζητήματα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Όσο προχωράμε λοιπόν στη δικιά μας Προεδρία με τους διάφορους φακέλους, κοιτούμε πώς να δημιουργήσουμε ένα σύστημα όπου οι διαφορετικοί φάκελοι μεταξύ τους έχουν συνοχή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεργάζονται διαφορετικοί εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με διαφορετικούς φακέλους, άρα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια πολύ καλή συνεργασία, όπως επίσης βέβαια και με τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. για παράδειγμα, και το είπε και η Επιτροπή, το θέμα των ε, εκπροσώπων και εκείνων που έχουν αναλάβει την φροντίδα των παιδιών. Πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό σύστημα όπου αναλαμβάνουμε έναν ανηλικά από τη στιγμή που κάνει αίτηση για άσυλο μέχρι να φτάσει στα 18 που δεν χρειάζεται πια κανένα κηδεμόνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη διαπιστώσει ότι υπάρχει μια μερική αντιμετώπιση από το Συμβούλιο. Μπορεί να φαίνεται αρνητικό εκ πρώτη όψεω, αλλά από την άλλη μεριά πρόκειται για ένα εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μα και το οποίο μα επιτρέπει τελικά να πετύχουμε αυτή τη συνοχή που θέλουμε. Για κάθε πρόταση λαμβάνουμε υπόψη μας τι αναφέρεται σχετικά στους άλλους φακέλους του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Δεν θέλουμε να προκαταλάβουμε δηλαδή τις συζητήσεις που θα γίνουν για άλλους φακέλους του πακέτου. Οπότε όλα αυτά διευκρινίζονται σιγά σιγά όσο ο κάθε φάκελος προχωράει και διαμορφώνεται όλο και περισσότερο. Έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσουμε καλύτερα να διασφαλίσουμε τη συνοχή ώστε σιγά σιγά να διαμορφωθεί και το τελικό αποτέλεσμα με συζητήσεις σε κάθε στάδιο. Για τον κανονισμό του Δουβλίνου τώρα, η Μαλτέζικη και η η Προεδρία έχουν κάνει ήδη πολύ σημαντικές προσπάθειες για να βγούμε από το αδιέξοδο όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Έγινε κάποια πρόοδος στις συζητήσεις και υπό τη δική μας Προεδρία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα για συμφωνία στο Συμβούλιο. Η Εστονική Προεδρία αναγνωρίζει βέβαια πόσο σημαντικό ήταν το καθήκον αυτό και πόσο δύσκολες ήταν οι συζητήσεις με όλες τις πλευρές, όλες τις χώρες μέλη. Εν μη τι άλλο τώρα καταλαβαίνουμε πού έγκυται τα προβλήματα, αλλά και πού μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος, κοινός παρονομαστής. Και ελπίζουμε σε αυτό που μένει από την Προεδρία μας να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τις χώρες μέλη, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου, που έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει συνένεση μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2018. Τώρα για την υπηρεσία σύλλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλω εδώ να μπω σε λεπτομέρειες για το που βρίσκεται αυτός ο φάκελος, το ακούσατε. Απλώς ελπίζουμε ως Προεδρία να καταφέρουμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών μας με το Κοινοβούλιο σύντομα στην Κορεπέρ για να τα εγκρίνει. Οπότε τα υπόλοιπα θα αποκλείονται από αυτή τη συμφωνία. Για την Eurodac, πρώτα απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα καλά αποτελέσματα στους τριμερείς διαλόγους. Για την Προεδρία μας είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε ακόμα όσο γίνεται περισσότερο μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες ουσιαστικά. Ακόμα κι αν για κάποια ζητήματα το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην έχει εντολή Ελπίζουμε παρόλα αυτά να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της ήδη υπάρχουσας ε, συμφωνίας. Για την αναδιατύπωση τώρα, ακούσατε ποια είναι η κατάσταση, αυτό που εμείς ελπίζουμε είναι ήδη την Τετάρτη μεθαύριο να μπορέσουμε να έχουμε εντολή για τριμερείς διαλόγους και να μπορέσουμε να αρχίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τριμερείς διαλόγους με το Κοινοβούλιο. Τώρα για την επανεγκατάσταση. Πράγματι την προηγούμενη εβδομάδα, 15 Νοεμβρίου, πιο σωστά, είχαμε εντολή για το Συμβούλιο και πολύ χαιρόμαστε που μπορούμε ήδη το Δεκέμβριο να έχουμε τον πρώτο τριμερή διάλογο. Και μετά θα συνεχιστούν βέβαια οι διαπραγματεύσεις και την επόμενη χρονιά. Για τον κανονισμό όσον αφορά τις δεξιότητες συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Αναφέρθηκε ότι η εντολή μας είναι μερική. Δεν έχουμε καταλήξει πουθενά. Όσον αφορά την εντολή ελπίζουμε ότι την Τετάρτη η εντολή θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο όσον αφορά την έννοια οικογενειακά μέλη. Οπότε θα έχουμε και περισσότερα να συζητήσουμε. στους δύο τελευταίους πολιτικούς τριμερείς διαλόγους και σε κάποιες άλλες συζητήσεις που θα γίνουν ελπίζουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο και να καταλήξουμε σε όσο γίνεται περισσότερα ζητήματα. Πάντως, πράγματι, χρειάζεται παραπάνω δουλειά που θα γίνει βέβαια υπό βουλγαρική προεδρία. Όσον αφορά τώρα τον κανονισμό για τις διαδικασίες ασύλου, είναι ένας περίπλοκος φάκελος αυτός και πολύ τεχνικός. Η πρώτη ανάγνωση οδήγησε στο να τελειώσουμε το Σεπτέμβριο. Οπότε αρχίσαμε αμέσως τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη ανάγνωση από πλευράς Προεδρίας τέλος πάντων και θα έχουμε τελειώσει τώρα αρχές Δεκεμβρίου πιστεύουμε με τη δεύτερη ανάγνωση, αλλά σίγουρα θα παραμείνει δουλειά και για τη συνέχεια. Δυστυχώς δεν θα έχουμε την εντολή για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο υπό τη δικιά μας Προεδρία. Αλλά προχωράει καλά αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι αυτά είναι όλα που είχα να πω εγώ. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Στόχος μας όμως ήταν να δουλέψουμε όσο γίνεται πιο σκληρά, να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο και να μην αφήσουμε τίποτα πίσω. Πρόεδρο, να μην αφήσετε τίποτα πίσω λέτε. Δύσκολο αυτό. Θα δούμε. Ανάλογα με τις δυσκολίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως δεν είναι εύκολη δουλειά αυτή. Είναι πολύ φάκελοι. Σας ακούσαμε προσεκτικά. Τώρα θα ακούσουμε τους εισηγητές. Ξέρω ότι τρεις η ώρα Δευτέρα μεσημέρι είναι δύσκολο να είναι όλοι εδώ, οπότε πολύ χαίρομαι που βλέπω εδώ τους εισηγητές. Λοιπόν, πείτε ό,τι έχετε να πείτε, θα έχετε χρόνο, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, με τη σειρά που ζητήσατε το λόγο. Η κυρία Σίπελ πρώτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα και την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ναι, τα θέματα είναι ευαίσθητα, είναι δύσκολα, είναι περίπλοκα. Υπάρχουν τόσες πολλές απόψεις. Τα ξέρουμε στο Κοινοβούλιο και ειδικά στην Επιτροπή μας. Αλλά με συγχωρείτε, εμείς καταλήξαμε σε μία θέση. Και τώρα, μετά από 18 μήνες, η Κομισιόν, και σας ευχαριστώ που το υπάρχουν τρία θέματα ακόμα, τρεις φάκελοι, που δεν υπάρχει θέση του Συμβουλίου. Τίποτα. Δεν μου λέτε λοιπόν ότι είναι δύσκολο. Το ξέρουμε, αλλά καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια θεση και τωρα μετα απο 18 μηνες ε, κομισιον και σας ευχαριστω που το υπαρχουν τρια θεματα ακομα τρεις φακελοι που δεν υπαρχει θεση του συμβουλιου τιποτα μην μου λετε λοιπον οτι ειναι δυσκολο το ξερουμε αλλα καταφεραμε να καταληξουμε σε μια θεση τωρα να συνεχίσω λέγοντας ότι αντιλαμβάνουμε ότι ειδικά το Συμβούλιο είναι έτοιμο να οριστικοποιήσει την ΕΑΖΟ, την Υπηρεσία Σύλλου και το ΓΥΡΟΝΤΑ. Καλά έχουμε δείξει ότι αν συμφωνήσουμε σε αυτά τα δύο θέματα, η όρεξη του Συμβουλίου να συνεχίσει να εργάζεται σοβαρά σε άλλα θέματα θα κοπεί ή δεν θα αυξηθεί να το πω έτσι, ταυτόχρονα για ε, επειδή ακριβώς ε, η φάκελη είναι δύσκολη και βεβαίως και εμείς εδώ μέσα είχαμε διαφορετικές θέσεις και μπορώ να σας πω και εγώ προσωπικά δεν είμαι ικανοποιημένη με όλα τα σημεία της συμφωνίας. Παρόλα αυτά, τώρα που έχουμε αυτές τις θέσεις, εμπιστεύομαι όλους τους εισηγητές εδώ στο Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά ότι θα παλέψουν για τις θέσεις ε, τις οποίες συμφωνήσαμε και πέρα από την γενική δήλωση ότι δεν βλέπω να αυξάνεται η όρεξη του Συμβουλίου για τα άλλα θέματα αν συμφωνήσουμε για την ΕΑΖΟ και τη Γιόντακ να πω ότι η ομάδα μου θα ήθελε να παλέψει για την θέση που βρήκαμε εδώ στο Κοινοβούλιο που αφορά παραδείγματο χάρη όχι μόνο τις περίοδους διατήρησης ε, κράτησης ε, και ας τα έχουμε αυτά κατά νου γιατί ίσως ε, το καλοκαίρι του 2018 της Βουλγαρικής Προεδρίας να έρθει μια πρόταση τι θα γίνει τότε, θα πάμε στις ευρωεκλογές και δεν θα υπάρχει ακόμα κάποια αλλαγή στην γενική πολιτική ασύλου. Και κύριε Πρόεδρε, μια πολιτική δήλωση θα ήθελα να κάνω. Ναι, γνωρίζω ότι δεν είναι ικανοποιημένα όλα τα κράτη-μέλη. Και νομίζω πως η Κομισιόν το είπε, ότι πρέπει οι Άζο και η Eurodac να σημειώσουν κάποια πρόοδο για να ικανοποιήσουν κάποια από τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε τελικά να έχουμε τη γενική αυτή μεταρρύθμιση. Αλλά να θυμόμαστε συμφωνήσαμε στην συμφωνία με την Τουρκία που είχε στόχο να κερδίσουμε λίγο χρόνο έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν και για το τι μπορούμε να κάνουμε με τρίτες χώρες και εσωτερικά. Δεν βλέπω λοιπόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εμείς λοιπόν κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Πρέπει να επιμείνουμε και να παλέψουμε για τις θέσεις μας και τώρα πρέπει να απαντήσει το Συμβούλιο γιατί δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια θέση για να διαπραγματευτούμε. Ευχαριστώ. Μάλιστα, αρχίσαμε βλέπω έτσι με ρυθμό. Να σας πω τώρα ποιοι θα είναι οι ομιλητές. Έχουμε ώρα. Για το Δουβλίνο, η κυρία Stevens και Wickstrom. Η κυρία Μπιόρκ για την επανεγκατάσταση, η κυρία Ίνετφελντ για τις συνθήκες υποδοχής, η κυρία Λάμπερτ. Κάποιος άλλος. Και η κυρία Γονμπέρκ. Κάποιος άλλος, όχι. Στίβενς, παρακαλώ. Hartelijk bedankt, voorzitter, beste collega's. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ακούσαμε πάρα πολλά για το καθεστώς κατάσταση. Προσπάθησε η Κομισιόν να δημιουργήσει ένα ενίο πλαίσιο μαζί με κάποιες συμφωνίες επανεισδοχής για να αυστηροποιηθεί η πολιτική της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο, το είδε κάπως αλλιώ τώρα, έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος θα υποχρεώνει δυστυχώς τα κράτη να δέχονται 100.000 ετούντες άσυλο το έτος και καταργείται το σκέλος των επιστροφών. Έχουμε αυτή τη συζήτηση στο πλαίσιο του κώδικα περί βίζας και είπαμε ότι δεν θα διαπραγματευτούμε περαιτέρω με αυτού του κειμένου και τώρα είναι στον κάδο των σκουπιδιών. Οπότε η ερώτησή μου είναι ποια είναι η άποψη των κρατών μελών για ένα τέτοιο μηχανισμό μετεγκατάστασης με κάποιους ελάχιστους όρους. Θα το συνδέσετε με το μηχανισμό βίζας. Σας ευχαριστώ. Ίσως ε, επειδή λείπα στην αρχή δεν τα ακούσατε όλα, αλλά φαντάζομαι θα σας ε, ενημερώσουν. Thank you, Chair, and thanks to all of you. I'd like to turn to my colleagues if there are some from my negotiating team. Θα ήθελα να ε, απευθυνθώ στους αδέλφους μου και να τους πω ότι σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνατε ε, και ιστορικό επίτευγμα πέντε πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούν πάνω από 200 και ακόμα της Ευρώπης συμφωνούν. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το ότι 28 όμως υπουργοί δεν μπόρεσαν τελικά να καταλήξουν σε μία και μόνο απόφαση. Εγώ θα τα λέω όλα αυτά μέχρι να υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου. Νομίζω ότι δουλέψαμε πάρα πολύ καλά όλοι μαζί και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και την υποστήριξη που δόθηκε ε, πριν από δύο εβδομάδες στην Ολομέλεια ε, όταν αμφισβητήθηκε η αρμοδιότητα της Επιτροπής μας και ήταν πολύ δύσκολη εκείνη η εποχή ε, δεχτήκαμε πίεση. Τώρα όμως έχουμε μια πλειοψηφία δύο τρίτων, ε, δηλαδή το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο με συντριπτική πλειοψηφία και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλω να επισημάνω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει επιτέλους να καταλήξουν σε κάποια θέση, να αναζητήσουν κάποια συμφωνία. Σύντομα θα μπούμε στο 18 και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε 14-15 μήνες όπου ε, θα μπορούμε ακόμα να διαπραγματευόμαστε για την νομοθεσία Τώρα, αν το Συμβούλιο σέρνεται ε, προσπαθώντας ε, να επιτύχει ομοφωνία για τη Συμφωνία του Δουβλίνου, ε, δεν θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις ή να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Και ξέρετε, φοβάμαι τελικά ότι κάποιοι το θέλουν αυτό, το επιθυμούν, θέλουν να συνεχίσουν να μας λένε ε, ότι είναι αδύνατο να καταλήξουμε σε κάποια θέση. Όμως ε, οι πολίτες ε, δεν αρέσκονται σε κάτι τέτοιο. Το 70% των πολιτών της Ευρώπης θέλουν η Ευρώπη να προσφέρει υπηρεσίε να τα καταφέρει σε θέματα μετανάστευσης. Κατανοώ βέβαια ότι αυτό δεν βολεύει το Συμβούλιο γιατί είναι πολύ πιο ευχάριστο για του υπουργού ε, κατά τη διάρκεια των συνδύσεών τους ε, να τα λένε χαλαρά από το να αναγκαστούν να βρουν κάποια ουσιαστική λύση σε ένα δύσκολο θέμα. Ε, δεν πρέπει όμως να υπάρχει μοφωνία. Να γιατί μπορεί και πρέπει να υπάρχει ειδική πλειοψηφία. Η Προεδρία αν έχει έστω κάποια πυγμή πρέπει να το υπογραμμίσει αυτό, ότι είναι αδύνατο να υπάρξει ομοφωνία. Υπάρχουν 4-5 χώρες που δεν θέλουν να γίνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν ξεχάστε την ομοφωνία και αρχίστε να αναζητάτε την πλειοψηφία. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στο Στρασβούργο την τελευταία φορά κατά την ψηφοφορία Εστονοί, Κροάτες, Βουλγάροι, ε, Ρουμάνοι, Λιθουανοί αυτοί ε, έδωσαν κατά δύο τρίτα υποστήριξη στην εντολή και στην πολωνική αντιπροσωπεία, ε, η Πολωνία που σήμερα είναι για να ντρεπόμαστε, εκεί το 50% των Πολωνών ψήφισαν υπέρ της εντολής και το 50% καταψήφισε. Έχω μπροστά μου τα ακριβή στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν να μην συνεχίσετε να ε, ονοματίζετε κρατημέλη. Πιστεύω ότι ακόμα και αν το Συμβούλιο δεν είναι τώρα έτοιμο για να κάνει αυτό το βήμα, θα πρέπει τουλάχιστον να αναζητήσει κάποια εντολή να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Πρέπει ειλικρινά να το σκεφτούν αυτό. Και ελπίζω ότι το Συμβούλιο μπορεί επίση να είναι λιγάκι και πιο ανοιχτό να προσπαθήσει να αναζητήσει κάποια έμπνευση ε, να αναζητήσει έμπνευση από τη δική μας θέση. Ξέρω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 ομάδες στο Συμβούλιο. Ίσως λοιπόν η δική μας η θέση να αποτελεί συμβιβασμό. Προσπαθήστε να το πουλήσετε ο συμβιβασμό και στο τέλος θα δείτε, θα είσαστε πολύ ευχαριστημένοι. Κατά την άποψή μου, όλες αυτές οι εκθέσεις για το κοινό ε, ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, εξαιρουμένη στις υπηρεσίες ασύλου, όλα αυτά πρέπει να προχωρήσουν ως δέσμοι διότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε ε, σε συμφωνία μόνο κάποιων τμήματων της συμφωνίας. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και επίσης δεν μπορούμε να δεχόμαστε το Συμβούλιο να δείχνει ότι θέλει να προχωρήσει μόνο σε κάποια τμήματα της δέσμης. Ε, τη γύροντα, ας πούμε, την θέλουν επαστησία, αλλά όχι τη Συμφωνία του Δουβλίνου και κάποια άλλα. Εγώ εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά είμαι επίση πεπισμένη ότι αν τελικά υπάρξει βούληση θα τα καταφέρουμε. Όμως η βούληση πρέπει να έρθει από το Συμβούλιο. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει πρέπει το Συμβουλίο να δείξει ε, κάποια ηγετική στάση και πολιτική βούληση. Αν δεν το κάνει η δουλειά μας πάει στράφη. Στη δημοκρατία κανείς ποτέ δεν μπορεί να είναι πάντα ευτυχισμένος. Αυτοί που κολυσιεργούν αν συνεχίσουν <clears throat> να προβάλλουν βέτο για τα πάντα, δεν θα πάμε πουθενά. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να ψηφίζουμε ε, με ειδική πλειοψηφία. Έτσι γίνεται σήμερα στην κοινωνία και αυτό να κάνει και το Συμβούλιο. Και αυτό πρέπει να το κάνει εχθές. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο και ελπίζω το Συμβούλιο σήμερα ε, να θέλει να ακούσει αλλά και να μεταφέρει περαιτέρω το μήνυμα ότι φτάνει πια μπουχτίσαμε, κουραστήκαμε. Ευχαριστώ. Σίγουρα θα μεταφέρει η Προεδρία το μήνυμα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Για την ε, επανεκατάσταση, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όντως, ε, η συνάδελφος ήταν απόλυτα σαφής και συμφωνώ κι εγώ. Είμαι όντω εισηγήτρια για την επανεγκατάσταση, οπότε και εγώ θέλω να αρχίσουν οι διαπραγματεύσει. 13 Δεκεμβρίου προβλέπεται. Αλλά εμείς το έχουμε πει από την ΚΟΕ ότι θέλουμε να δουλέψουμε για αυτό το θέμα ως πακέτο. Το θέλουμε αυτό το πακέτο ασύλου και θέλουμε συνοχή. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσει. Αν λοιπόν κατακαιρματίσουμε τους διάφορους φακέλους, θα αποτύχουμε και δεν θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτών που μας εξέλεξαν να έρθουμε εδώ. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει συνοχή. Και για το Δουβλίνο δεν βλέπω να προχωράμε. Η Σεσίλια τα είπε και εμείς συμφωνούμε και ανησυχούμε όλος ιδιαίτερος. Και όταν μιλάω για συνοχή, το ακούμε συχνά συνοχή, συνοχή, συνοχή, αλλά δεν νομίζω ότι το Συμβούλιο έχει συνοχή. Εμείς ναι, είπαμε ότι που θα έχουμε ένα σύστημα ή που δεν θα έχουμε ένα σύστημα. Ενώ το Συμβούλιο λέει θα προχωρήσουμε τους φακέλους που έχουν περισσότερη σημασία και θεωρεί ότι είναι συνοχή. Για μας δεν είναι αυτό συνοχή, όχι δεν θέλουμε να προχωρήσουμε μόνο για το Γιούρντά ή για δεν ξέρω τι. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια και βλέπω ότι εκεί προχωρούν ε, σύντομα και γρήγορα. Καμιά φορά συνατιόμαστε στις 10 η ώρα το βράδυ. Ναι, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του αυτό. Δεν συμφωνώ με τέτοιου είδου διαδικασίε. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν συμφωνώ με τέτοιε διαδικασίε. Το Συμβούλιο θέλει να προχωρήσει ένα φάκελο, τον ε, προχωράει, αλλά μένει πίσω στα άλλα. Όχι, δεν συμφωνούμε με μια τέτοια διαδικασία. Οπότε, περιμένω και εγώ να προχωρήσει και στους άλλους φακέλους στο Συμβούλιο για να μπορέσουν όλα να λειτουργήσουν και να μπορέσει να λειτουργήσει και ικανοποιητικά το σύστημα στο σύνολό του. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Σαφέστατο το μήνυμά σας. Η Σοφή Χετφέλ τώρα που είναι υπεύθυνη για τον φάκελο που αναφέρεται στην υποδοχή. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσείς ε, βεβαίως είστε απλώς οι αγγελιοφόροι και υπηρετείτε τους ε, νότερους σας, αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω πλήρως με τις τρεις προλαλήσεις σας. Και αυτό το οποίο μου προξενεί εντύπωση είναι η τεράστια αντίθεση μεταξύ των της πολύ πολύ πολύ αργής ή καθόλου ουσιαστικά πρόοδου στις επίσημες πολιτικές σύλλου και την απίστευτη ταχύτητα με την οποία το Συμβουλίο κλείνει συμφωνίες με δικτάτορας και άλλα τέτοια έτσι, περίεργα καθιστώτα. Η λεγόμενη δήλωση με την Τουρκία έκλεισε μία νυχτή και περιμένουμε μία θέση του Συμβουλίου ναι, αυτό το θέμα 1,5 χρόνο. Είναι λίγο περίεργο δηλαδή. Αποφασίζουν να ξοδέψουν δισεκατομμύρια ευρώ σε αποτυχημένα κράτη και δικτατορίες και αυταρχικά καθεστώτα χωρίς κανένα πρόβλημα και δεν μπορείτε να προχωρήσετε στο θέμα του ασύλου σε μια πολιτική ασύλου που υπάρχει έτσι απλά αρνούνται να την ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη και αυτό το οποίο κάνουμε εδώ πέρα είναι να βελτιώνουμε το σύστημα και να ελπίζουμε μετά ότι τα κράτη-μέλη θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί παραβιάζουν τις συνθήκες αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη. Παραβιάζουν τις συνθήκες, δεν ακολουθούν την πολιτική ασύλου και παριστάνουν ότι εξακολουθεί να ισχύει η ομοφωνία. Δεν λέει αυτό η συνθήκη. και επίσης ε, βεβαίω απογοητεύεται τους πολίτες γιατί όπως είπε η Σεσίλια Βίξτρομ ο κόσμος ε, θέλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελέσματα. Λοιπόν, Κοινοβούλιο και Κομισιόν έχουν αποτελέσματα. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ποιο φταίει. Οι κυβερνήσει. εγκαταλείπουν τους Ευρωπαίου πολίτε, γιατί, γιατί φοβούνται τους ψηφοφόρους. Α, ξέρετε κάτι. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών θέλει να καλωσορίσει τους πρόσφυγες και μετανάστες. Δύο πράγματα θέλουν να ξέρουν. Πρώτον, ότι μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση και ξέρετε κάτι ναι μπορούμε. Είμαστε, έχω πει ξανά, η πιο πλούσια Ήπειρος στον πλανήτη, πάνω 500 εκατομμύρια άνθρωποι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, ναι, μπορούμε. Και δεύτερον, θέλουν να γνωρίζουν ότι η αύξηση των μεταναστών δεν θα επηρεάσει καθόλου τις δικές τους ευκαιρίες και δικαιώματα. Έχουν ε, βεβαίω ε, δικαίωμα. Ε, αλλά οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να φροντίσουν ότι έχουν προσβάσεις σε δουλειές, υγεία, εκπαίδευση κτλ. Εντάξει, ας σταματήσουμε λοιπόν εδώ πέρα. γιατί βλέπω ότι τα κράτη-μέλη εδώ πέρα βραδιπορούν, αλλά ότι είναι εξωτερική ανάθεση τρέχει. Ευρώπη, Φρούριο κτλ. Όχι, είναι παροδία. Δεν είναι αλήθεια. Η ε, Ευρώπη, Φρούριο δεν ισχύει. Ασχοληθείτε λοιπόν με το να προωθήσετε τα ζητήματα που είναι επιτάπητος και βρείτε μια αποτελεσματική πολιτική ασύλου που θα ευθυγραμμίζεται και με τις αρχές μας. Και τέλος, για την προσέγγιση πακέτο, συμφωνώ με τους άλλους εισηγητές, θα το ψηφίσουμε ως πακέτο και να τα ξεκαθαρίσω, πακέτο δεν σημαίνει ευθυγράμμιση προς τα κάτω, σημαίνει ότι θα έχουμε μια πολιτική ασύλου αποτελεσματική και ανθρώπινη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ βεβαίω ε, με πολλά από αυτά τα οποία ακούστηκαν. Προσπαθώ έτσι να αποκτήσω μια εικόνα της όλης διαδικασίας, μια αίσθηση του τι θέλουν τα κράτη-μέλη τελικά. Και νομίζω ότι ε, δεν είναι σαφές. Ναι, υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν, αλλά όπως είπε η Σόφη, αυτό δεν σημαίνει ότι θα οπισθοχωρούμε. Είναι συναρπαστικό ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να τόσα, τόσες ρήτρες που είναι ίσως και μήπως κτλ σε έναν κανονισμό. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι κάτι το οποίο ναι θα βελτιώσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη αλλά και την κατάσταση για τους ετούντες άσυλο. Και έχω άρα μια ερώτηση για το εάν υπάρχει συνοχή και για το εάν τα κράτη-μέλη ε, ποινικοποιούν τις ε, δευτερογενείς μετακινήσεις ή ε, λένε ότι ο κόσμος θα πρέπει να παραμείνει που είναι αλλάζοντας ε, το Δουβλίνο και βεβαίως με το να μην υπάρχει μια απόδοση του συστήματος η οποία θα ήταν κίνητρο να μετακινηθεί ο κόσμος. Με ενδιαφέρει λοιπόν το κατά πόσον νιώθουν τα κράτη-μέλη μια αίσθηση αλληλεγγύης στην ε, χρηστή διοίκηση. Γιατί βεβαίως ε, το θέμα είναι το, ότι, το πώς βλέπουμε το θέμα των ασυνόδευτων λύκων λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά γνωρίζουμε ότι οι επιχειρησιακές πτυχές ε, των όσων έχουμε είναι πραγματικά απέσιες. Και πολλοί νέοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να μετακινούνται δεν μετακινούνται γιατί τα κράτη-μέλη ε, δεν συνεννοούνται και δεν είμαι πεπισμένη ότι το να δώσουμε περισσότερες ευθύνες στην ΕΑΖΟ ενώ δεν ξέρουμε ακόμα ποιες θα είναι οι αλλαγές είναι κάτι το σωστό. Γνωρίζουμε, όπως ανέφερε η Κομισιόν, ότι θα απαιτηθούν περισσότεροι πόροι. Γνωρίζουμε ότι δεν έχουν προϋπολογιστεί και επίσης είναι δύσκολο να ζητήσουμε σοβαρές αλλαγές εκεί, εάν δεν είναι σαφές το ποια θα είναι μετά η νομοθεσία. Και όσον αφορά την ελληνική μεταξύ κρατών μελών, θα ήθελα να ακούσω από το Συμβούλιο εάν θεωρούν ότι αυξάνεται η αλληλεγγύη ή ότι έχουμε ακόμα κάποια κράτη-μέλη αμετακίνητα που δεν θέλουν να επιδείξουν αλληλεγγύη. Δεν θέλουν να υπάρξει ένα γενικό σύστημα και ε, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ποια είναι αυτά, αλλά εάν αν ισχύει αυτό να γίνει πιο σαφές για να συνεννοηθούμε με τους συναδέλφους μας για να αλλάξουμε την κατάσταση. Όπως είπα λοιπόν, ε, υπάρχουν μέλη που αναγνωρίζουν ότι κάποιοι επιτόπου ε, είναι διατεθειμένοι να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Σούιμπερκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση, αλλά πρέπει να σας πω ότι τώρα έχω πιο πολλά ερωτηματικά από πριν. Πολλά χρήζουν διευκρίνησης. Αναφέρθηκε ότι πρόκειται για θέματα πολιτικά, σημαντικά, πράγματι ε, και στα κράτη-μέλη ε, το θέμα της ε, αναγκαστικής κατανομής αυτό θα είναι θέμα που θα μας απασχολήσει και σε επόμενες εκλογές. Ε, υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα που δεν μπορούν να επιληθούν και αυτά είναι τα εξή. Ναι, εναρμόνιση στις προϋποθέσεις και τις απαιτήσει, αλλά ποιο κράτος μέλος θα εκλειφθεί όσο μέσο όρο. όρος, η Ρουμανία ή η Σουηδία. Η διάσταση μεταξύ των δύο είναι τεράστια. Μετά, Δουβλίνο 5, ανακατανομή. Αναφέρθηκε ότι όταν θα έχετε επιτευχθεί ένα ανώτατο όριο, ε, θα πρέπει να λαμβάνει ε, κάποιο άλλο κράτος. Εμείς ε, έχουμε πάρει πολλούς ασύλους, ετούντες άσυλος στη Σουδία, και αναμένουμε και τις οικογένειές τους. Αυτό τώρα θα ληφθεί υπόψη ή θα αγνοηθούν οι οικογένειες. Υποτίθεται 80.000 πρέπει να επιστραφούν πίσω. Αυτό δεν το καταφέρνουμε μόνοι μας. Ζητήσαμε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα ερωτήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Αυτά είχα να σας πω από δικής μου πλευράς. Και μετά, όσον αφορά στα κονδύλια, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λένε ότι τα κράτη-μέλη που δεν δέχονται πρόσφυγες θα πρέπει να τιμωρηθούν οικονομικά. Αν όμως αποφασίσουν ορισμένα κράτη-μέλη να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το έχετε λάβει υπόψη σας. Υπάρχουν 7-8 κράτη που δεν θέλουν να πάρουν πρόσφυγες. Ε, σας έχει απασχολήσει αυτό. Ε, για να δούμε τι θα γίνει όταν η Βουλγαρία θα αναλάβει την Προεδρία. Θα τα παρακολουθώ όλα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Πριν ε, λοιπόν δώσω το λόγο στον ε, εκπρόσωπο της Εστονικής Προεδρίας, νομίζω ότι Ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Δεν θα μπει η Προεδρία σε λεπτομέρειες, δεν θα ονοματίσει συγκεκριμένες χώρες, να μην είμαστε υπερβολικοί στις προσδοκίες μας, αλλά νομίζω ότι ένα πράγμα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Μίλησαν όλοι οι συγητές, αλλά νομίζω και ο εισηγητής για τις απαιτήσει θα πει ακριβώς το ίδιο, ότι είναι μια, ένα πακέτο, μια δέσμη μέτρων. Αυτή είναι η προσέγγιση. Όσον αφορά την υπηρεσία και τη Eurodank, νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Υπάρχει και διάσταση απόψεων στην Επιτροπή. Όμως δέσμη, το πακέτο πρέπει να παραμείνει, δεν πρέπει να κατέβουν οι απαιτήσει. Για να δούμε τι θα γίνει. Πώς θα τα καταφέρει η Εστονική Προεδρία. Μπορεί να επιφέρει ρήξη. Δεν πιστεύω, αλλά λέμε. Ίσως ε, μπορούμε να εκπέμψουμε ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τη Συμφωνία του Δουβλίνου, ε, η δέσμη μέτρων δεν πρέπει να μειώσει τις ε, απαιτήσει. Πολλοί από εμάς έχουμε κάνει την εμπειρία των ε, πακέτων για το άσυλο στην τελευταία θητεία και την καταστροφή που ακολούθησε. Εάν λοιπόν τα κρατημέλη ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία θα υπάρξει πρόβλημα εμπιστοσύνη από πλευράς πολιτών. Εγώ λοιπόν απλά επισημαίνω τη σοβαρότητα της δουλειάς των συναδέλφων. Ίσως ε, το Συμβούλιο μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά που επισήμανα και ίσως μπορεί και κάποιος άλλος ε, ε, να τοποθετηθεί. Νομίζω όμως ε, ότι όλα είναι απόλυτα σαφή. Ίσως μπορείτε να τοποθετηθεί τουλάχιστον σε αυτά που είπαν οι συγητές. Ο κύριος Ράιαν. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους τους συζητητές για τις παρεμβάσεις τους. Το γενικό μήνυμα το ακούσαμε σαφώς. Καταλάβαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα βλέπει όλα αυτά τα θέματα ως πακέτο. Βέβαια διαστάθηκα κύριος από τον κυρία Βίλστρομ κάποιο άνοιγμα ότι ίσως η κατάσταση με τη νέα εντολή για την υπηρεσία μπορεί να είναι κάτι που θα δούμε λίγο διαφορετικά. Η Επιτροπή το ενθαρρύνει αυτό. Θέλω επίση να υπογραμμίσω ότι το ωφέλη που πιστεύουμε ότι θα πορεύουν από την εντολή τη υπηρεσία θα έχει μια μόνιμη αξία που θα αντιληφθούμε πολύ σύντομα. Γιατί θα υπάρχει η λειτουργική στήριξη που θα μπορεί να δίνει η υπηρεσία στι χώρε μέλη εξαιτία των πόρων που θα έχει στη διάθεσή τη, τι αρμοδιότητες που θα αναλάβει την ε, ελεγκτική της λειτουργία θα φροντίσει δηλαδή να εφαρμόσουν οι χώρες μέλη την νομοθεσία έτσι ως έχει. Για το πακέτο, εντάξει, το καταλάβαμε. Έχω και μία παρατήρηση. για αυτό που είπατε πολλοί από εσά ότι δηλαδή η συνθήκη προβλέπει ψηφοφορία με πλειοψηφία, οπότε εδώ τίθεται το ζήτημα χρειάζεται ή όχι συμφωνεί όλων. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πολιτικός, οπότε δεν θέλω να μπω σε άλλα χωράφια έξω από αυτά της Επιτροπής, αλλά νομίζω ότι εξή τον κόπο εδώ να πούμε, ότι δεν εκπλήσει το γεγονός ότι για ένα θέμα τόσο βασικό, υπαρξιακή σημασία θα έλεγα σχεδόν, εννοείται ότι γίνεται κάθε προσπάθεια από πλευράς του Συμβουλίου για να προσπαθήσει να πετύχει συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών είναι σαφές. Για να μπορεί να είναι βιώσιμη όποια απόφαση παρθεί τελικά και να μπορεί να λειτουργήσει, έχει νόημα να προσπαθήσουμε να πετύχουμε όσο γίνεται ευρύτερη συνένεση στο Συμβούλιο. Οπότε με αυτή την έννοια δεν εκπλήσει το γεγονός ότι κρατάει καιρό και ότι είναι δύσκολο. Μπορεί να είναι προφανές, αλλά παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι καλά κάνουμε και το υπογραμμίζουμε ξανά και ξανά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Και το τελευταίο μου, για αυτά που είπε η κυρία Λάμπερτ. για τα ανάμεικτα μηνύματα που έρχονται από τις χώρες μέλη όσον αφορά τις ε, προδιαγραφές και την φιλοδοξία εναρμόνισης. Είναι αλήθεια. Αλλά έχουμε δει και είναι θετικό. Αποδοχή σε ένα βαθμό από τις χώρες μέλη για αυξημένη εναρμόνιση. Δεν είναι ένα συμπέρασμα που ισχύει για όλα και πάντα, αλλά υπάρχει μια τέτοια στάση των χωρών μελών που έχει αλλάξει σε σχέση με το πώς ήταν πριν από 18 μήνες. Υπάρχει μια αποδοχή της ε, Ενισχυμένη εναρμόνισης. Πολύ περισσότερο τέλο πάντων σήμερα από ό,τι κατά το παρελθόν. σε ευχαριστούμε. Αυτό που λέτε δηλαδή είναι ότι προσπαθείτε να βοηθήσετε, ότι το Συμβούλιο προσπαθεί να πετύχει ε, συνένεση. Και αν σας καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία επειδή το θέμα είναι τόσο πολύ σημαντικό. Αυτό προσπαθείτε να μας πείτε. Γιατί αν προσπαθείτε να πετύχετε συνένεση από τις χώρες μέλη σε αυτό το ζήτημα, θα είμαστε εδώ μέχρι τον επόμενο αιώνα. Η ευελιξία, νέος τρόπος σκέψης. Αυτά δεν χρειάζονται. Δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, εντάξει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφώς και αναγνωρίζει τι προβλέπουν οι συνθήκες για την έγκριση νομοθεσίας. Με ειδική πλειοψηφία δηλαδή. Αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να πετύχουμε συμφωνία με τρόπο που, πώς να το πω, να διχάζει όσο γίνεται λιγότερο τους εμπλεκόμενους. Γι' αυτό λέω ότι γίνεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί ευρεία συνένεση, όσο γίνεται πιο ευρεία. Είναι φυσιολογικό. Ακριβώς επειδή είναι τόσο ευαίσθητο αυτό το ζήτημα. Ε, προφανώς και η φιλοδοξία του Συμβουλίου είναι αυτή να πετύχει όσο γίνεται ευρύτερη συνένεση και αυτό πολεμάει. Πρόεδρος, εντάξει, το κατάλαβα. Δεν εκπλήσει, αλλά είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να αλλάξει κάπως ο τρόπος σχέσης και σκέψης και να πετύχουμε κάποιες επιμέρους συμφωνίες, αλλιώς τι θα γίνει. Η κυρία Σίπελ θέλει διαδικαστικό. Όχι, όχι, πρόεδρε, μία πρόταση μόνο θέλω να πω. Ναι, θα μπορούσα να συμφωνήσω ότι αξίζει να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλες τις χώρες μέλη να συμφωνήσουν. Ε, το κάναμε με το σημερινό πακέτο ασύλου το οποίο δεν εφαρμόζεται. Οπότε για μένα το επιχείρημα αυτό που λέτε δεν ισχύει. Πρόεδρος, ναι, ναι, γι' αυτό κι εγώ βλέπετε ότι διστάζω να συμφωνήσω μαζί σας. Γιατί έχουμε βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση σήμερα που... Ναι, λέτε ότι δεν εφαρμόζεται. Ναι, μερικές χώρες δεν το εφαρμόσουν καθόλου. Ίσως αυτό είναι η συνέπεια ότι όλοι βιάστηκαν να συμφωνήσουμε κάτι που ξέραν ότι δεν θα εφαρμόσουν. <clears throat> Εν πάση Το βασικό είναι ψηφοφορία και απόφαση με πλειοψηφία. Σε αυτό πρέπει να προχωρήσουμε. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να βοηθήσετε και να βρείτε τρόπους να συμφωνήσουν όσο γίνεται περισσότεροι. Ωραία. Τώρα. Προεδρία. Η κυρία Λούς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για όλες αυτές τις παρεμβάσεις που ακούσαμε από τις χώρες μέλη. Ε, συγγνώμη, από τους ευρωβουλευτές. Υπάρχει κάτι εδώ που πρέπει να διορθώσω. Σήμερα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη φορά το Συμβούλιο, ποτέ δεν υπόθηκε ότι θέλουμε να βγάλουμε από το πακέτο είτε τη Eurodac είτε οτιδήποτε άλλο Ούτε η Επιτροπή είπε κάτι τέτοιο, ούτε το Συμβούλιο συζητάει κάτι τέτοιο. Αυτό θέλω να το διορθώσω, έτσι. Να μην ε, μείνουμε με παρεξήγηση. Όμως, δουλεύοντας πάνω σε όλους αυτούς τους φακέλους εδώ και μήνες, ναι, πράγματι, κάποιοι φακελοί προχωρούν πιο γρήγορα. Κάποια θέματα, ε, για κάποια θέματα πετυχαίνουμε πιο γρήγορα συμφωνία από ό,τι για άλλα δεν είναι θέμα στρατηγικής να ολοκληρώσουμε το ένα ή το άλλο. Όχι, στόχος της προεδρία μας είναι να προχωρήσουμε με όλους τους φακέλους και με το Δουβλίνο, να πετύχουμε σε βιβασμούς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οπότε, ναι, κάποιοι φάκελοι είναι πιο περίπλοκοι, πιο δύσκολη συμφωνία για αυτούς. Και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς γιατί έχουμε και το EPR. Όλα αυτά εκεί καταλήγουν. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, με, προχωράμε από 27 διαφορετικά, 28 διαφορετικά συστήματα και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο να λειτουργεί. Και πού μπαίνουν οι προδιαγραφές. Ποια είναι προδιαγραφές θα ακολουθήσουμε. Είναι δύσκολο. Οπότε αν την Τετάρτη πετύχουμε εντολή, θα γίνει ακόμα πολλή δουλειά. Και ήδη έχει γίνει πολλή δουλειά που πρέπει να συνεχιστεί. μπορούμε να προχωρήσουμε καλά. Γι' αυτό και ειλικρινά ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το δικό σας το έργο που ήταν πολύ καλό Δεν είναι θέμα στρατηγικής μας να προχωρήσουμε στον ένα φάκελο και όχι στο, σε κάποιον άλλο. Και κάποια ακόμα σχόλια. Ρωτήσατε κατά πόσο το Συμβούλιο θέλει να καταλήξει σε μια κατάσταση όπου η Επιτροπή να αναγκαστή να αποσύρει την πρότασή της. Όχι! Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα έχουμε πολυάριθμες συναντήσεις. Γίνονται πολλά. Και έχει επιτευχθεί πρόοδος, που είναι σημαντική. Χρειάζεται βέβαια κι άλλη. Είναι αλήθεια, αλλά έπρεπε να γίνουν αυτά που έγιναν. Μην κοιτάμε μόνο τι μένει να γίνει. Ας δούμε και τι έχει γίνει και μέχρι τώρα. Οπότε, ειδικά για να λειτουργήσουν στην πράξη όσα θέλουμε να αποφασίσουμε. Κοιτάξτε, οι προτάσεις της Επιτροπής, ε, συγγνώμη που το λέω, δεν ήταν ε, τέλειες. Υπήρξε συνέπεια που έπρεπε να διορθωθεί αυτά για το θεματικό και αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε τώρα. Και για να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο να μπορέσει να λειτουργήσει και να καταλαβαίνουν και οι χώρες μέλη τι κάνουν και τι αποφασίζουν, όλοι τις χρειαζόμαστε αυτές τις συζητήσεις. Παίρνουν χρόνο και είναι δύσκολες, αλλά είναι για να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα στο τέλος, πιο ανθρώπινο, πιο αποτελεσματικό, που είναι προς όφελος όλων. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε χρόνο. Δουλεύουμε συνέχεια και γίνεται πρόοδος. Μην το παραβλέπετε κι αυτό. Πρόοδος. Αυτό με σοκάρει, είπατε ότι δεν ήταν τέλειος όλες οι προτάσεις της Κομισιόν. Εγώ είμαι εδώ ανέκαθεν. Δεν φταίει η Προεδρία, το ξέρουμε. Φταίνει οι χώρες μέλη όταν προχωράει ένας φάκελος δεν προχωράνε άλλοι. Εντάξει, εσείς έχετε επομιστεί όλο το βάρος, εσείς πρέπει να συντονίσετε τις χώρες μέλη, εσείς τα ακούτε. Τέλος πάντων, ξέρουμε ότι υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Είμαστε συνομοθέτες. Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά τις τεχνικές δυσκολίες που έχουν σαν αποτέλεσμα ένας φάκελος να προχωρά πιο γρήγορα, ένας άλλος λιγότερο. Υπάρχουν διαρθρωτικοί λόγοι, ναι, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Η κυρία Λάμπερτς είχε κάνει για, την πρώτη, για τον πρώτο οργανισμό. Τα ξέρουμε, ναι. Να είμαστε σαφείς. Στείλαμε τα πολιτικά μας μηνύματα, τα οποία θα πρέπει να περάσουν όσο έγιναν. Τα έκαναν οι εισηγητέ και είμαι γνώμων που τα είπαν έτσι όπως τα είπαν ξεκάθαρα. Ας ελπίσουμε να προχωρήσουμε και με τις εντολές γρήγορα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συζητητές για τη σκληρή τους δουλειά. Και αυτοί και το προσωπικό τους και η γραμματεία ε, δουλεύουν τόσο σκληρά όσο δεν νομίζω να έχω δει ποτέ να δουλεύουμε τόσο σκληρά στην Επιτροπή μας. Και η Προεδρία σίγουρα το ίδιο και το προσωπικό της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε επεξεργαστεί πολλούς φακέλους και κατά το παρελθόν. Αλλά αυτή τη φορά πραγματικά. Μπράβο και σας ευχαριστώ. Ό,τι πολιτικό μήνυμα όμως σας μεταφέραμε, ελπίζουμε να περάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν συνάδελφοι για το πακέτο αυτό και την Επιτροπή και την Προεδρία. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στο σημείο 4. Διαδικασία επιπαραβάση κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Συνάδελφοι, επειδή ε, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, καθυστερήσαμε λίγο ε, μέχρι να έρθουν οι συνάδελφοι, ε, θα ξεκινήσουμε τώρα το επόμενο θέμα, το οποίο αφορά την διαδικασία παραβάση για την ελευθερή μετακίνηση. Για να σας δώσω μια γρήγορη εξήγηση. Στις 25 Σεπτεμβρίου ζητήσαμε Ζητήσαμε την Κομισιόν να έρθει εδώ να συζητήσουμε ένα γραπτό ερώτημα που υπέβαλαν διάφοροι βουλευτέ για την διαδικασία παραβάση βάρου του ΕΒ Βασιλείου για την εφαρμογή τη οδηγία περί ελεύθερη μετακίνηση, ε, ζητήματα τα οποία δεν είχαν απαντηθεί εγκαίρω. Σύμφωνα με το άρθρο 130 παραγραφος 4 λοιπόν του κανονισμού, η Κομισιόν οφείλει να έρθει ενώπιον της Επιτροπής μας ε, για να απαντήσει. Τα μέλη της ΛΥΜΠΕ θεώρησαν ότι η απάντηση που δόθηκε δεν ήταν ικανοποιητική και προτάθηκε να ζητήσουμε από την Επιτροπό Γιούροβα περισσότερες πληροφορίες. κυρία Γιούροβα κολλείεται σήμερα, αλλά η κυρία Μαρή Ελέν Μπούλανζε επικεφαλής της ε, σχετικής, ε, του σχετικού τμήματος Κομισιών, θα μας ενημερώσει. Έχετε τον λόγο λοιπόν. Κυρία Μπουλάνζε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν είμαι ακόμα σε θέση να πω εάν η Κομισιόν θα προσφύγει στο δικαστήριο για το δικαίωμα διαμονής οικονομικά μη ενεργών πολιτών και το ζήτημα του εάν η σχέση με το NHS μπορεί να θεωρηθεί ασφάλιση υγείας. Θα ήθελα ως αφετηρία να πω πως το αίτημα οι μη οικονομικά ενεργοί πολίτες να έχουν ασφάλιση υγείας προβλέπεται από την Οδηγία Ελεύθερης Μετακίνησης στο αρθρο 7.1.Β. Το σημείο απόκλησης με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το εάν η ασφάλιση στο NHS θεωρείται συνολική ασφάλιση υγείας ή εάν οι μη οικονομικά ενεργοί πολίτες απαιτείται να έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Η Κομισιόν ακόμα αξιολογεί την περίπτωση. Γνωρίζω ότι θεωρείται ότι καθυστερούμε Παρ' όλα αυτά επιτρέψατε μου να τονίσω ότι για να μπορέσουμε να πάμε στο δικαστήριο πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τα επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Αυτό απαιτεί δυστυχώς ε, περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα σε τρία σημεία. Τις διαδικασίες, ε, το πολιτικό πλαίσιο και την ουσία επί της διαδικασίας θα ήθελα να τονίσω ότι η παράβαση αυτή είναι μέλος ενός ευρύτερου φακέλου που αφορά το κατά πόσον συμμορφώνεται το Βρετανικό Δίκαιο με την οδηγία περί ελευθερής μετακίνησης. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με την περίπτωση 2011 2.0 αφορούν πάνω από 100 περιπτώσεις συμμόρφωσης ε, που ε, θίξαμε με τις Βρετανικές Αρχές από όταν ετέθη η σχετική οδηγία. Συγκεκριμένα από το 2009 η Κομισιόν ξεκίνησε 27 πιλωτικές έρευνες θέμης για την εφαρμογή του δικαιώματος ελεύθερη μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. να πούμε ότι οι καταγγελίες ε, πολιτών είναι 1,4 ε, των σχετικών καταγγελιών που λαμβάνει η Κομισιόν. Είναι ένα περίπλοκο θέμα ε, το οποίο απασχολεί την Κομισιόν και είμαστε σε τακτική επαφή με τις Βρετανικές Αρχές. Η Κομισιόν έχει κάνει πολλά βήματα για να σημειωθεί κάποια πρόοδος. Η πρόοδος των ερευνών της Κομισιόν όσον αφορά το θέμα της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου από το Ηνωμένο Βασίλειο είχε επίσης, ε, είχαν επίσης επηρεαστεί και από την συνεργασία με τις Βρετανικές Αρχές. Και εδώ πέρα θα ήθελα να έρθω στο πολιτικό πλαίσιο, ότι πρόκειται για μια δυναμική και εξελισσόμενη υπόθεση. Από όταν ετέθη ενισχύ η σχετική οδηγία τον Απρίλιο του 2006 και, άρχισε, και μεταφέρθηκε στο Βρετανικό Δίκαιο, το Ηνωμένο Βασίλειο τροποποίησε 19 φορές ε, την σχετική νομοθεσία, μία μισή φορά κάθε χρόνο δηλαδή και 9, 11 με τροποποίησης έγιναν από όταν ξεκίνησε η διαδικασία επί παραβάση, δηλαδή δύο τροποποιήσεις το έτος. Η αλλαγή του νόμου βεβαίως ε, συνοδεύτηκε και με διαφορετικές εγκυκλίους ε, προς το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών και όπως γνωρίζετε οι εγκύκλοι αυτοί είναι πολύ σημαντικές στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάση. Από όταν ξεκίνησε η διαδικασία, το δικαστήριο έβγαλε πέντε αποφάσεις που ερμηνεύουν τον σχετικό κανονισμό και αφορούν τους όρους που θα πρέπει να ισχύουν σε σχέση με το δικαίωμα εγκατάστασης των μη οικονομικά ενεργών πολιτών και την ασφαλής υγείας και μία στην ε, επιστροφή υπηκών. Οι αποφάσεις αυτές ε, έχουν ζητήσει να αξιολογηθεί εις βάθος η νομική κατάσταση σε σχέση με αυτό και να αναφέρουμε ότι η περίπτωση αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εξεταστεί εντελεχώς στο εσωτερικό της Κομισιόν μετά την απόφαση του δικαστηρίου οι αρμόδιες υπηρεσίες Κομισιόν συναντήθηκαν τακτικά για το θέμα αυτό και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Επί τη ουσίας τώρα στο τρίτο μέρο. Η Κομισιόν πρέπει βεβαίω να, είναι, να πατά πολύ γερά στα πόδια της από νομική σκοπιά και θα πρέπει ακριβώς να δούμε το ζήτημα πρόσβασης οικονομικά μη ενεργών πολιτών σε κάποια επιδόματα. Ανέφερα και κάποιες περιπτώσει σε περίπτωση Ιντάνο, Αλιμάνοβιτς, Γκαρσιανέτο και την μια περίπτωση που χάσαμε και την περίπτωση Γκούζα που εκρεμεί. Όπως είπαμε, η Κομισιόν έχασε την υπόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο αντίκτυπος λοιπόν της πρόσφατης αυτής νομολογίας μπορούμε να πούμε ότι είναι ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να αρνηθούν να δώσουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας στους μη ενεργά οικονομικού πολιτές. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα άτομα αυτά δεν θα εμποδίζονται από το να εκπληρώσουν τους όρους για να έχουν δικαίωμα κατοικίε για πέρα από τρει μήνες. Δηλαδή, κυρίως τον όρο του να έχουν ασφάλιση υγείας. Για το λόγο αυτό, οι μετακινούμενοι πολιτέ θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συνεισφέρουν αναλογικά σε κάποιο σύστημα ασφάλισης υγείας ε, στο κράτος συνήθως κατοικία τους. Για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, παρά το ότι θεωρούμε ότι η ασφάλιση του NHS δεν είναι συνολική ασφάλιση υγείας, οι οικονομικά ανενεργοί ε, πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν δωρεάν θεραπεία από το NHS με βάση την Βρετανική νομοθεσία. Καθώς λοιπόν δεν ε, υπάρχει ανάγκη να καταγραφούν κάπου στο Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρούν ότι κατοικούν νομίμως στη χώρα επειδή μέσω της σχέσης τους με το NHS ε, έχουν ασφάλιση υγείας. Πρέπει λοιπόν αυτή η αντίφαση να απαντηθεί οριστικά. Και για να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου θα ήθελα να αναφερθώ στην θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στις διαπραγματεύσεις για το άρθρο 50 και στο εγγραφό θέσεων του Ιουνίου 2017 και στην τελευταία δημοσίευση διοικητικών διαδικασιών του Νοεμβρίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο λέει ότι δεν θα απαιτήσει στοιχεία και αποδείξεις ότι οι οικονομικά ανενεργοί πολίτες είχαν ασφάλεια υγείας στο παρελθόν για να, για θεωρεί ότι ε, είχαν συνεχή κατοικία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βιντεβέλη ε, Σοφή <clears throat> έχει το λόγο. Τα άκουσα όλα αυτά και προσπάθησα λιγάκι να φανταστώ Πώς αισθάνεται κανείς όταν είναι πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και παίρνει μια επιστολή που του λένε ότι ε, θα απελαθείς ε, από τη χώρα γιατί δεν καλύπτεις τις ε, προδιαγραφές αυτής της σχετικής οδηγίας που συζητάμε. Πώς αισθάνονται κανείς ακούγοντας αυτά που είπε η σας. Δηλαδή ε, να αναγκαστεί κανείς ε, να ε, φύγει από την οικογένειά του, να χάσει το σπίτι του, να χάσει τη σύνταξή του και να πάρει αυτή την, επιτροπή, την απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατανοώ ε, κύριε Πρόεδρε, ότι η κυρία Μπουλαντζέ είναι απλά ο αγγελιαφόρος ε, και δεν πρέπει να σκοτώνουμε τον αγγελιαφόρο, αλλά η συζήτηση έχει ξαναγίνει. Μας είπατε τότε και καταλήξαμε ότι η απάντηση θα πρέπει να δοθεί σε πολιτικό επίπεδο. Και πού είναι η Επιτροπή. Εντάξει, κατανοώ ότι η Επίτροπος ε, είναι ιδιαίτερα αποσχολημένη, αλλά μιλάμε για 3,3 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να τους εξυπηρετήσουν ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και συγγνώμη τώρα αυτή την απάντηση μας δίνεται. Μιλάμε για ανθρώπους ε, οι οποίοι έχουν υπαρξιακή αγωνία για το μέλλον τους. Και θα είχε την καλοσύνη η να με ακούσει, αν δεν σας πειράζει. Ειλικρινά, αυτά που μας είπατε, δεν ξέρω τι να πω, έχω μείνει εννοεί. Ε, ξεκίνησε διαδικασία επί παραβάση το 2012 πριν από πέντε χρόνια και μας λέτε ότι εξακολουθείτε να κάνετε έρευνες και μάλιστα ε, και το φταίξιμο ε, στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου γιατί αλλάζει συνεχώ ε, του νόμου. Συμφωνώ μαζί σα ότι η χάλια είναι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά δεν είναι αυτό δικαιολογία. Εσεί πρέπει να εφαρμόζετε τον νόμο. Η Επιτροπή πρέπει να κάνει τη δουλειά τη. Και ειλικρινά θα ερευνήσω το ε, κατά πόσον μπορούμε να στείλουμε την Επιτροπή στα δικαστήρια για παράληψη καθήκοντος, γιατί πραγματικά δεν υπηρετείτε τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που πληρώνουν το μισθό σας, το δικό σας, εσείς που είστε εκεί. Συγγνώμη πρόεδρε, αλλά μιλάμε για κανονικούς ανθρώπους με κανονικές ζωές που ε, κινδυνεύει η ύπαρξή τους και η ζωή τους ε, και σας ρωτώ εσάς τι θα κάνει το Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε συνεχώς να λέμε τα ίδια πραγματικά είμαι εξοργισμένη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν κάνει τίποτα, παραλείπει να δράσει. Και ρωτώ πρώτα, τι θα κάνουμε τώρα. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε, ότι πράγματι αυτή είναι η δεύτερη συζήτηση για το θέμα αυτό και είχα καλέσει την Επίτροπο να έρθει εδώ. Σωστά τα λέτε τα γεγονότα, ότι είχαμε καταλήξει το θέμα να ανέβει σε πολιτικό επίπεδο. Σωστό αυτό ως ε, στοιχείο για να το ξέρουν και άλλοι συνάδελφοι. Τελικά δεν ήρθε βέβαια η Επίτροπο, σωστό και αυτό. Η κυρία Λάμπερτ. Ναι, καταλαβαίνω την ε, απογοήτευση και την οργή όλων. Εδώ συμβαίνουν πολλά και διάφορα πράγματα συγχρόνως. Πρώτα απ' όλα, οι κανόνες αλλάζουν, αργούν οι απαντήσεις από τις χώρες μέλη. Ξέρουμε ότι υποφελούνται κιόλας από αυτό και αποφεύγουν άμα δεν θέλουν να απαντήσουν. Όμως υπάρχει και το θέμα πολιτικής απόφασης που υπάρχει όχι μόνο για αυτό, αλλά και για άλλα ζητήματα. Η Επιτροπή κάνει πίσω, αντί, αντίθετα να ορμήσει περισσότερο, γιατί επειδή πριν υπήρχε το δημοψήφισμα, μετά είχαμε τα αποτελέσματα του δημοψήφισματος και το καθεξής. Εμείς όμως είμαστε πολιτικοί, αυτό είναι ένα πράγμα. Ο κόσμος όμως αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες. Το θέμα της υποχρεωτικής ασφάλισης για το Ενωμένο Βασίλειο, όχι μόνο, αλλά κυρίως είναι από τα πράγματα τα οποία αγχώνουν πάρα πολύ τον κόσμο. Ακριβώς επειδή αλλάζουν οι κανόνες χωρίς να ενημερώνεται ο κόσμος ή το χωρίς να ενημερώνεται όπως θα έπρεπε. Αυτό είναι Κάτι που το ξέρουμε γιατί έρχεται ο κόσμος και μας βρίσκει. Τι κάνεις όταν έχουν αλλάξει οι κανόνες αλλά δεν σε έχουν ενημερώσει επαρκώς ή δεν είναι αρκετά σαφείς οι αλλαγές στις ιστοσελίδες κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να εκφράσει στην Επιτροπή την ανησυχία μας εξαιτία της έλλειψης δράσης. Καταλαβαίνω ότι θέλω να κάνω τα πράγματα καλά, καταλαβαίνω ένα σώρο δυσκολίες, εντάξει, αλλά αν είχαμε προχωρήσει νωρίτερα, νομίζω ότι εκεί θα είχαμε δείξει τι θέλουμε και θα είχαμε βοηθήσει τον κόσμο και στον Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αλλού. Στον Ηνωμένο δημιουργείται βέβαια ένα μεγάλο πρόβλημα επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να βγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να ξέρετε το θέμα της οδηγίας για την ελεύθερη διακίνηση κολλάει και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες χώρες. Κάθε φορά λοιπόν που δεν ε, δρούμε, που κάνουμε πίσω, όπως η Επιτροπή σε αυτή την περίπτωση, είναι ένα πολύ κακό μήνυμα που στέλνουμε και είναι σε βάρος των πολιτών μας. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και τις δύο για ό,τι είπατε. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι αν δημιουργείται εδώ αίσθηση και τα λέει κανείς έξω από τα δόντια, καταλαβαίνετε γιατί έτσι. Ήταν σωστή για το πολιτικό επίπεδο, κυρία Χετβέλτ. Η απάντηση που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτό που μπορούμε να έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι το πολιτικό. Και ίσως τους συντονιστές. Όχι εγώ, αν το βάλει κάποιος συντονιστής, είπε η κυρία Λάμπερτς ότι πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει. Ωραία, να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό βάσει της σημασίας που αξίζει το ζήτημα, έτσι. Νομίζω ότι οι ευρωβουλευτές πάντως το είπαν ξεκάθαρα το τι συμβαίνει και το τι περιμένουμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά θα το θέσουμε, είπαμε, στην επόμενη συνάντηση συντονιστών. Εντάξει. Σόφη, θες να προσθέσεις κάτι. Ναι, Εντάξει, συντονιστέ. Ωραία. Ό,τι και να γίνει όμω, μπορούμε να το κάνουμε γρήγορα. Είναι 1,5 χρόνο που έχει περάσει. Δεν γίνεται, ο κόσμο δεν μπορεί να περιμένει. Μην περιμένουμε ακόμα εβδομάδε και μήνε. Ωραία. στι 6 Δεκεμβρίου θα το βάλουμε στι συνεδρίε των συντονιστών. Έτσι και θα φροντίσουν να ενημερωθούν όλοι για τις λεπτομέρειες. Θα το βάλουμε για τις 6 του μηνός. Εντάξει. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε για αυτό το θέμα. Θα το θέσουμε, είπαμε, στην επόμενη συνεδρία συντονιστών. Λοιπόν, έχω τριμερή διάλογο που πρέπει να πάω. Η κυρία Γκάλ συμφώνησε να με αντικαταστήσει εδώ στο Προεδρείο για τα επόμενα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Καλησπέρα σα, συνάδελφοι. Προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. για την παρουσίαση της κατάστασης ε, του τρεμερούς διαλόγου για το θέμα, για το θέμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, πιστοποιήσεων ταξιδιού αιτίας. Θα ήθελα να πω δύο λόγια πριν δώσω τον λόγο στους συναδέλφους. Ε, πρέπει να γνωρίζετε ότι πρόταση, η Κομισιόν παρουσίασε μία πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών επιβατών τον Νοέμβριο του 2016. Η Κομισιόν ψήφισε στις 19 Οκτωβρίου τη θέση του Κοινοβουλίου και μου δόθηκε η εντολή στην επόμενη όλο ολομέλεια για να ξεκινήσω τι διαπραγματεύσει με το Κομισιόν Συμβούλιο. Από όταν επιβεβαιώθηκε η εντολή, είχαμε τριμερείς διαλόγους ε, τον Οκτώβριο και στις 16 Νοεμβρίου και θα έχουμε και την Τετάρτη άλλο ένα γύρο. Οι διαλογοί αποδεικνύουν ότι οι συνομοθέτες ε, γνωρίζουν την ε, σημασία του θέματος ε, και την προτεραιότητα που έχει και εξέφρασαν ε, διάθεσή να βρεθούν κάποιες συμβαστικές λύσεις. Θα ήθελα τώρα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για την συμμετοχή τους στο θέμα αυτό και στους τριμερείς διαλόγους. Επιπλέον είχαμε έξι συναντήσεις στο τεχνικό επίπεδο με τους συμβούλους και τους βοηθούς μας ε, και την Κομισιόν και το Συμβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βοηθούς μας και τους συμβούλους μας ε, για την εξαιρετική και κουραστική δουλειά που έκαναν. Αυτό το οποίο βλέπουμε μέχρι στιγμής καθώς ε, αυτή τη στιγμή υπερασπίζουμε ξεκάθαρα τις προτάσεις μας και προσπαθούμε να εξηγήσουμε τις θέσεις μας γιατί ξέρετε ότι ε, το Συμβούλιο ε, επιμένει στην θέση του και το Εκομισιόν έχει κάποιες καλές ιδέες για συμβιβασμό. Τα πιο προβληματικά ζητήματα μέχρι στιγμής είναι η περίληψη των επιβατών transit, το εάν το ΕΤΙΑΣ θα πρέπει να θεωρείται όρος εισόδου και παραμονής ή μόνο εισόδου, ε, το Συμβούλιο Δεοντολογίας του ΕΤΙΑΣ και τι μορφή θα έχει, εξαιρέσεις από το ΕΤΙΑΣ και η διατήρηση δεδομένων. Ελπίζω λοιπόν να βρεθούν ε, καλές συμβαστικές λύσεις Τώρα, εμείς ε, θεωρώ ότι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την θέση μας ε, και τα σημαντικότερα σημεία που είχαμε μέχρι τώρα στο έργο της Επιτροπής, ε, θεωρώ ότι πρέπει να ισχύσουν τρεις αρχές. Το ένα είναι ότι με την αίτιας δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε χειρότερους όρους από ό,τι όταν ζητάει κανείς βίζα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να είναι χειρότερο Προσπάθησα επίσης ε, το ΕΤΙΑΣ να έχει ε, συνάφεια με το σύστημα εισόδου-εξόδου και βεβαίω με το ΔΙΣ ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να ζητάει λιγότερα και οπωσδήποτε όχι περισσότερα. Και τέλος δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε υπερβολικά τον μηχανισμό έτσι ώστε να μην ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είμαστε λοιπόν ακόμα στην αρχή της αναζήτησης συμβιβαστικών προτάσεων. Έχουμε νομίζω καλό κλίμα και ελπίζω να συνεχίσουμε και να έχουμε μια συμβαστική λύση η οποία σημαίνει ότι κανείς δεν θα είναι ικανοποιημένος. Ελπίζω λοιπόν όταν έχουμε κάποιε βελτιώσεις ε, να μπορέσω να έρθω να σας πω ότι έχουμε και καλά νέα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ε, κυρία Συγήτρια, σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ όλους όσοι δούλεψαν πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά πολύ μου αρέσει πώς το δουλεύουμε. Ακόμα και αν στην ομάδα μου διαφωνούμε θεμελιωδώς με το ζήτημα. Εξακολουθώ να λυπούμε που βιαζόμαστε να εγκρίνουμε το κείμενο αυτό, γνωρίζοντας ότι πριν από το 2020 δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Οπότε θα μπορούσαμε να πάρουμε μερικούς μήνες παραπάνω για να καθίσουμε σοβαρά να δουλέψουμε, αντί να βιαζόμαστε για κάτι το οποίο έτσι κι δεν θα μπορέσει να δουλέψει τώρα. Φαίνεται ότι όλοι θέλουν πριν τη λήξη της Προεδρίας αυτής να το έχουμε τελειώσει το θέμα. Γιατί το νέο σύστημα αυτό αίτια, το ευρωπαϊκό σύστημα δηλαδή πληροφοριών και αδείας ε, ταξιδίου, είναι κάτι ε, τοπικό. Εγώ το ονομάζω μάλιστα τοπική θεώρηση, βίζα. Λέτε ότι με τίποτα το σύστημα αυτό δεν πρέπει να καταλήξει να ζητάει πράγματα τα οποία δεν ε, ζητάμε από κάποιον που χρειάζεται θεώρηση. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τα, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Τα περισσότερα δεδομένα, έτσι κι αλλιώς, εδώ βασίζονται σε δήλωση. Οπότε δεν βλέπω σε τι μας διασφαλίζει το να ζητάμε από κάποιον να κάνει επιπλέον δηλώσεις. Το μόνο που κάνουμε έτσι είναι να συσσωρεύουμε παραπάνω δεδομένα. Και έπειτα εκπλήσωμε και με τη θέση του Συμβουλίου με την οποία συμφωνεί και η Επιτροπή, ενώ στην αρχή δεν ήταν έτσι, για τους ε, επιβάτες transit. Γιατί έτσι θα ζητάμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και όπως πολύ σωστά είπατε, θα αποθαρρύνουμε κάποιους ανθρώπους να περνάνε transit από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν χρησιμοποιώ συνήθως οικονομικά στοιχεία, αλλά εδώ μου φαίνεται τόσο παράλογο οικονομικά που ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Όταν ε, ζητάμε όλα αυτά ε, που θέλουμε να ζητήσουμε από αεροπορικές ε, εταιρείες και μάλιστα από αυτές που βρίσκονται σε πιο εύθραυστη θέση. Εμείς λοιπόν στην ΚΟΕ θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε επί της ουσίας πάνω στο κείμενο αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά κι άλλο, ώστε το κείμενο αυτό να είναι όσο γίνεται πιο λογικό στο τέλος. Νομίζω ότι μερικοί παραλογίζονται εδώ όσον αφορά την συλλογή δεδομένων. Θέλουν να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη, αλλά δεν καθησυχάζουν τους πολίτες, γιατί όλα αυτά τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τίποτα άλλο παρά μόνο για να βάζουν τον κόσμο που τα δίνει σε μια κατάσταση ανασφάλειας ακριβώς, γιατί ανησυχούν για το πώς θα χρησιμοποιηθούν, αν θα είναι αναλογική χρήση τους, αν θα χρησιμοποιηθούν για λόγους για τους οποίους δεν προβλέπονται κλπ. Και για το θέμα του transit, νομίζω ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρέπει να εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμόστε για τα υπόλοιπα, τουλάχιστον για τους ε, επιβάτες transit πρέπει να ισχύει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Βερζιά. Αν δεν θέλει κανείς άλλος το λόγο, τότε θα συνοψίσω λέγοντας ότι συμφωνούμε με πολλά από αυτά που ακούστηκαν. Φυσικά και έχουμε διαφορές, αλλά προς το παρόν η δουλειά έχει προχωρήσει καλά, με καλή συνεργασία και ελπίζω ότι έτσι θα συνεχίσουμε. Ο τριμερής διάλογος ο επόμενος την Τετάρτη θα δείξει αν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς και ελπίζουμε να μας βοηθήσει με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι και γι' αυτό. Και περνάμε στο επόμενο θέμα. Είναι αξιολόγηση της απειλής που αντιπροσωπεύει το οργανώμενο έγκλημα <clears throat> στο διαδίκτυο. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ευρήματα όσον αφορά τις απειλές από το οργανωμένο έγκλημα στο κυβερνοχώρο και έχει να κάνει βέβαια και με τους ρυθμιστές και με τους πολιτικούς κλπ. Ο κύριος Φιλίπα Μαν που είναι προστάμενος της Μονάδας Στρατηγικής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στο Κυβερνοχώρο της Europol είναι μαζί μας εξετάζουμε εδώ πέρα τι συμβαίνει και ρυθμιστικά αλλά και στην σκοτεινή πλευρά όπως τη λέμε. Ευχαριστώ κύριε Μάν που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σας δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Δέκα λεπτά παρακαλώ. Μετά θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Παρακαλώ. Thank you, Mrs. Chair, and uh, thank you, members of the Committee. Ευχαριστώ πολύ τα μέλη της Επιτροπής που μου δίνει τη δυνατότητα να σας ε, παρουσιάσουμε την απαρχίδα των προγραμμάτων μας. Ε, την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Εκείνο λοιπόν που καθιστά την έκθεση αυτή κάπως μοναδική είναι ότι ε, προσφέρει και τη δυνατότητα εφαρμογής του νόμου για θέματα ποινική δικαιοσύνης. όλα αυτά στηρίζονται και από τον κλάδο γενικότερα. Είναι μια πολύ περιεκτική έκθεση η οποία όχι μόνο εξετάζει τις προκλήσεις σε κάποιο βαθμό προσπαθεί και να προβλέψει το μέλλον και αυτό που έχει σημασία είναι και ότι προσφέρει μια σειρά συστάσεων σε εκείνους που λαμβάνουν αποφάσεις, που επιβάλλουν τον νόμο αλλά και που χαράσουν και πολιτική. Έχουμε λοιπόν μια διαρθρωμένη διαδικασία για να αποκτάμε πληροφορίες. Την ε, αναλύουμε, ε, έχουμε έρευνες, συνεντεύξεις ε, σε ακαδημαϊκούς φορείς, σε πάρα πολλούς χώρους. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Τώρα, ας δούμε ποια είναι τα θέματα που καλύπτονται στην έκθεση. Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία σε τρεις τομείς. Είναι αντιμετώπιση της κακοποίησης των ανηλίκων, το έγκλημα με χρήση υψηλής τεχνολογίας, αλλά κοιτάμε και άλλα θέματα ε, όπως οι επιθέσεις κατά της υποδομής, οι προκλήσεις από το Internet of Things, ε, προκλήσεις που έχουν σχέση με τα big data, αλλά και ε, θέματα που έχουν σχέση με τον κυβέρνο χώρο. Σε αυτή την έκθεση υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Αυτή η έκθεση είναι και δημόσια τώρα, είναι δημοσιοποιημένη. το 2014 πρώτο ξεκινήσαμε, δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο και υπάρχει τώρα πλέον στην ιστοσελίδα μας. Επιπρόσθετα από τα θέματα αυτά έχουμε και άλλα πιο εξωτικά. Παραδείγματο χάρη πέρυσι εξετάσαμε ε, θέματα κρυπτογραφημένα. Η κρυπτογράφηση ε, αυτό το είχαμε δει και κατά το παρελθόν σε σχέση με την ε, τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομπατική, ε, πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν την, τα θέματα που σχετίζονται με την επιβολή του νόμου. Ή τους hackers και αυτά τα εξετάζουμε κάτω από το δικό μας πρίσμα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από πλευράς επιβολής του νόμου για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Αν τώρα ε, πρέπει να επιλέξω δύο πράγματα από τη φετινή έκθεση, θα είναι το Mirai Botnet. Αυτή η ονομασία χρησιμοποιήθηκε πέρυσι ε, για να ε, μπορούμε να περιγράψουμε συσκευές, κάμερες που μετατράπηκαν σε κακοπροαίρετα εργαλεία από εγκληματίες και με τον τρόπο αυτό υπήρξε καταγραφή στοιχείων που βοήθησαν σε επιθέσεις. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν τώρα είναι κάτι το οποίο είχε προβλεφθεί κατά το παρελθόν, αλλά είναι η πρώτη χρονιά ε, που οι εγκληματίες χρησιμοποιούν ως όπλα συσκευές μη ασφαλείς. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό στην οθόνη σας, αλλά αν έχετε πληγεί από κάποιον ιό, θα έχετε δει αυτή την οθόνη, ίσως ε, αυτό να προέκυψε τυχαία, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικό. Αυτό προέκυψε το Μάιο του 2017. Είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα για το τι μπορεί να συμβεί αν συνδυάσει κανείς ε, διάφορα στοιχεία ε, και συμπεριλάβει και το στοιχείο το τυχαίο. Αυτό το είχαμε και ε, μετά από τρεις μήνες είχαμε πράγματι μία επίθεση δεν τα λέω αυτά από το μυαλό μου. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν κάποιες βασικές απειλές. είναι το τυχαίο με το επαναλαμβανόμενο και αυτό πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη απειλή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν. Αυτά τώρα είναι μια γενική εικόνα των βασικών τάσεων και απειλών όπως τις έχουμε καταγράψει. Αυτά είναι κάτω από το πρίσμα της αστυνομία. Πολλά από αυτά που βλέπετε είναι ε, αυτά που αναφέρονται στις αστυνομικές ε, αρχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις ε, αυτά είναι διαφορετικά ε, από αυτά ε, που τα κατανοούν και τα γνωρίζουν οι ακαδημαϊκοί. Το ransomware ε, είναι μια πολύ σημαντική απειλή, ε, θα συνεχίσει να υπάρχει, έχει σχέση με το Internet of Things, γιατί έχουμε όλο και περισσότερες συσκευές ε, που συνδέονται στο διαδίκτυο και αυτές θα μπορούν να είναι ο στόχος μιας επίθεσης ransomware. με συντηρητικέ αξιολογήσεις ε, θα έχουμε πολύ σύντομα περίπου 20 δισεκατομμύρια συσκευέ που θα συνδέουν το διαδίκτυο. Άλλοι μιλάνε για 100 δις συσκευές. Ε, καταλαβαίνετε ότι οι ανησυχίες επιτείνονται και θα ξέρετε φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα. Ε, ίσως πρέπει να συζητήσουμε για τους κατασκευαστές αυτών των συσκευών, αλλά οι συσκευές ήδη υπάρχουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να δει κανείς λιγάκι την υποδομή. Όσον αφορά την κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών. Αυτό έχει άμεση σχέση και με τον ε, εξαναγκασμό και την εκμετάλλευση των ε, παιδιών. Ε, σχετικά με την παραβίαση των δεδομένων, δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει αυτό. Έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα τέτοιες παραβιάσεις που έλαβαν χώρα για να προκύψουν εγκλήματα. Η κατάχρηση του dark web σχετικά με, τη, με το dark web ε, δεν είναι μόνο μία απειλή αλλά στηρίζονται και πάρα πολλές ε, μορφές ε, εγκλημάτων. Αυτό που βλέπουμε με τη νέα τεχνολογία που πλέον παρουσιάζεται στην αγορά είναι ότι οι εγκληματίες βλέπουν αυτή τη νέα τεχνολογία, το πώς μπορούν να κάνουν κατάχρηση αυτής αλλάζουν τα μοντέλα, οι εγκληματίες προσαρμόζονται στη νέα τεχνολογία, σε νέες δυνατότητες και αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι αστυνομικές αρχές, οι αρμόδιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδράσουν σε κακόβουλες πράξεις. Παράδειγμα, πέρυσι είχαμε επιτυχημένη δράση ε, κατά το Expert Kit Market που το χρησιμοποιούν εγκληματίε ε, για επίθεση κατά των υπολογιστών. Αποτέλεσμα αυτού το Expert Kit Market σε μεγάλο βαθμό εξαφανίστηκε και οι εγκληματίε ε, πλέον χρησιμοποίησαν άλλες τακτικές και το spam ε, υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. εξακολουθεί να υπάρχουν, εξακολουθούν να υπάρχουν και απάτες ε, σε σχέση με τις ε, πιστοτικές ε, κάρτες. Αυτό εξακολουθεί να υφίσταται. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται Μιλάμε, μιλήσαμε για το ransomware, ε, το οποίο θα εξακολουθήσει να είναι ε, μία από τις πιο σημαντικές ε, κακόβουλες πράξεις και απειλές μιλήσαμε για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τον εξαναγκασμό που έχει σχέση με τα παιδιά. Βλέπουμε ότι οι δράστες σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε εργαλεία που ξαναγκάζουν μάλλον τα παιδιά να τα χρησιμοποιήσουν. Οι εγκληματίες ε, λοιπόν ε, κάνουν κατάχρηση όπως σας είπα πολλών εργαλείων. Ε, κυρίως όσον αφορά την ε, παιδική πορνογραφία, οι ε, δράστες, ε, οι αυτούργοι έχουν πολύ ψηλά πρότυπα και επίπεδα ασφαλείας. Σχετικά τώρα, νομίζω ότι έχω αναφέρει, ήδη τι σαπάτες με τις κάρτες, ο ηλεκτρονικός τομέας πωλήσεων έχει πληγεί πάρα πολύ οι απάτες με τις κάρτες εξακολουθούν να υπάρχουν ε, διότι ε, δεν εφαρμόζονται οι απαραίτητες προδιαγραφές. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Έχουμε λοιπόν το σκοτεινό δίκτυο, τις σκοτεινές αγορές. Είναι μια απειλή που αφορά πολλούς τομείς ε, εγκλημάτων όχι μόνο το κυβερνό έγκλημα, αλλά και πολλά παραδοσιακά εγκλήματα, θα τα χαρακτήριζα όπως ε, το εμπόριο ναρκωτικών, ε, λατρεμπόριο όπλων, ε, παραποιημένα και παραχαραγμένα έγγραφα και το καθεξής. Επόμενη διαφάνεια. έχουμε επίσης ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιούν οι εγκληματίες ακόμα και στην περίπτωση πολύ ε, πολύπλοκών επιθέσεων. Συχνά ε, το πρώτο βήμα είναι μια κοινωνική επαφή, η κοινωνική μηχανική όπως λέμε. Γιατί είναι ευκολότερο βεβαίως να παρακάμψουμε τους, ε, τα ανθρώπινα εμπόδια παρά τα τεχνολογικά. Και έχουμε και τις απαντήσεις που αναφέραμε πριν, δηλαδή αλλαγές στην συμπεριφορά των διοκτικών αρχών και των εταιριών και εξακολουθούν άρα να βασίζονται σε αυτά τα μέσα οι εγκληματίες. Και πάλι βεβαίως τα κρυπτονομίσματα, ειδικά το bitcoin γιατί έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, αλλά βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν και άλλα κρυπτονομίσματα τα οποία παρέχουν ένα μεγαλύτερο βαθμό ανωνυμίας και προστασίας. Επόμενη διαφάνεια. για να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπαμε για τα μοντέλα εγκληματικότητας. Ξεκινώντας από το 2014, αυτό το οποίο περιγράψαμε ως μια βιομηχανοποίηση του κυβερνού εγκλήματος. Δηλαδή, για να διαπράξει κανείς ε, το κυβερνό έγκλημα, μπορεί να αγοράσει τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που απαιτούνται γι' αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε το έγκλημα ως υπηρεσία η οποία παρέχεται σε άλλους εγκληματίες. Οπότε όταν μιλάμε βέβαια για την ε, κυβερνοτρομοκρατία είναι μια μεγάλη μας ανησυχία και έχουμε κάποια εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα για, ε, σε διάφορους εγκληματίες. Επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα μια εικόνα των νομικών και τεχνικών προκλήσεων που αντιμετωπίσουμε στην έρευνα και δίωξη του κυβερνοεγκλήματος. Ε, γενικό είναι αυτό το οποίο βλέπετε. Έχουμε έξι τίτλους οι οποίοι βεβαίως ε, υποκρύπτουν πολύ συγκεκριμένες προκλήσεις. Έχουμε την εγκληματική χρήση της κρυπτογράφησης, ε, οι ζητήματα πολιτικής, οι προβλήματα, αν θέλετε, στην υποδομή του διαδικτύου που διευκολύνουν τους εγκληματίες των χρησιμοποιήσουν την υφιστάμενη τεχνολογία. Επίσης η απώλεια της τοποθεσίας, η ανώνυμα δίκτυα όπως το TOR ε, επίσης σχετίζονται με το cloud computing και τα σχετικά νομικά ζητήματα. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ούτε καν εντός τη Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ε, κοινό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του κυβερνού εγκλήματο που σχετίζεται σε έναν βαθμό και με την διεθνή συνεργασία. Όλοι γνωρίζετε τις προκλήσεις γύρω από την διαδικασία ΕΜΛΑΤ και το πόσο δύσκολο είναι να ζητάμε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία από τρίτες χώρες. Οπότε όταν μιλάμε για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος οποιοδήποτε εγκλήματος πια, γιατί όλα έχουν ένα τέτοιο σκέλος, πρέπει να συνεργαστούμε με τον κλάδο και με άλλους ε, εταίρους. Και το πρόβλημα εκεί είναι ότι δεν υπάρχει ένα τυποποιημένο πλαίσιο του τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να μοιραστούμε κτλ. Και τέλος, κάτι το οποίο αφορά ειδικά τις διοκτικές αρχές είναι το πώς ε, δημιουργούμε ακριβώς ε, τις ε, δεξιότητες για να καταπολεμήσουμε το κυβερνό έγκλημα και τις απειλές που υπάρχουν στον κυβερνοχώρο και πώς τις διατηρούμε βεβαίως αυτές τις δεξιότητες. Επόμενη διαφάνεια. Ε, δεν είναι λοιπόν όλα τα πράγματα όπως είπαμε σκοτεινά έχουμε κάποιες βασικές συστάσεις, κλειδιά, πράγματα τα οποία μπορούμε να κοιτάξουμε για να βελτιώσουμε την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με την πρόληψη και την ενημέρωση. Το καλύτερο απ' όλα είναι να προλαμβάνουμε ένα έγκλημα αντί να το διερευνούμε εκ των υστέρων και έχουμε πολύ επιτυχίες εκστρατείες πρόληψης η καμπάνια πείτε όχι το οποίο αφορά ειδικά τον σεξουαλικό εκβιασμό και εξαναγκασμό βασίζεται σε μια έκθεση εδώ πέρα των διοκτικών αρχών αλλά και μια διαβάθμιτη έκθεση η οποία δόθηκε στο κοινό είναι κάποια βίντεο υψηλής ποιότητας και στο τέλος κάθε βίντεο βλέπουμε το σημείο επαφή για την κάθε ώρα π.χ. Ολλανδία, Γερμανία κτλ. Για τη συγκεκριμένη χώρα δηλαδή θα έχουμε το που μπορεί κανείς να είναι σε επαφή αν έχει πέσει θύμα τέτοιου εγκλήματος. Το άλλο θέμα ανέφερα το σκοτεινό και το βαθύ δίκτυο ως ε, βασικές προκλήσεις. Εκεί πέρα λοιπόν προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με τους εταίρους μας, διοπτικές αρχές ε, και τις εταιρείε για να έχουμε μια κοινή στρατηγική προσέγγιση για να δούμε το έγκλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε με μια πιο στρατηγική προσέγγιση για να δούμε την εγκληματικότητα στον κύβερνο χώρο, αλλά όπως είπαμε και οι εγκληματίες είναι αρκετά ευέλικτοι. Μια άλλη σύσταση που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε ακριβώς το έγκλημα ως υπηρεσία, πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτούς οι οποίοι παρέχουν τα ε, εργαλεία, κλίδια της υπηρεσίας αυτές. Και μετά, τελευταίο, ε, να τονίσουμε το ότι χρειαζόμαστε πιο επαρκή νομοθεσία, κάτι το οποίο μπορεί να είναι και μεταφορά της υφιστάμενης νομοθεσίας στο εθνικό επίπεδο για να έχουμε μια αναλογική και αποτελεσματική αντίδραση στο κυβέρνο έγκλημα. Αλλά το βασικό είναι η συνεργασία, συντονισμός όλων των σχετικών εταίρων με τρόπο ώστε να προλάβουμε τις ε, καταστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Δύο βουλευτές έχουμε εδώ, την κυρία Στίβενς και τον κύριο Άλμπρεχτ. Ε, Η κυρία Στίβενς πρώτη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαν. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε για να μας παρουσιάσετε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα στο διαδίκτυο. Να αρχίσω πάλι από την αρχή, μια που βάλατε τώρα τα ακουστικά σας. Ωραία, θα αρχίσω και πάλι από την αρχή. Λοιπόν, έλεγα, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αμών που ήρθε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε για να μας παρουσιάσετε την κατάσταση όσον αφορά την εγκληματικότητα online στην Ευρωπαϊκή Ένωση σας ρωτάω ως συνεισηγήτρια, επειδή μιλάμε συχνά για τις μεγάλες επιχειρήσεις ε, δεδομένων, για να αποφύγουμε πώς ε, μπορεί να προχωρήσει η προπαγάνδα που γίνεται online, για παράδειγμα για το τζιχαντισμό. Εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει. και πώς αυτό συνδυάζεται με την ελευθερία έκφρασης. Και τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτού. Ζητώ συγγνώμη που για οικογενειακού λόγους θα πρέπει να φύγω. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Και σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ βρίσκομαι. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Είναι πολύ σημαντικό το έργο σας. Και ελπίζω να έχουμε και άλλες ευκαιρίες να ανταλλάσσουμε απόψεις για όλες αυτές τις προκλήσεις. Εγώ σε ένα θέμα θα επικεντρωθώ και για το οποίο θέλω να έχω τις απόψεις σας και τα σχολιά σας. τη δυνατότητα. Πώς μπορούμε να έχουμε στοιχεία από επιχειρήσεις είτε που δεν εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε που αποθηκεύουν τα δεδομένα του αλλού, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται συζήτηση, εμπλέκεται και η Europol και οι αρχές των χωρών μελών, για αυτήν ακριβώς την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Είτε γιατί οι επιχειρήσει μας έχουν την έδρα τους ε, αλλού, είτε αποθηκεύουν αλλού τα δεδομένα τους, χωρίς δηλαδή να περνάμε από την ε, κανονική διαδικασία. που έχει να κάνει με τρίτες χώρες. Οπότε ρωτάω, πιστεύετε ότι εδώ υπάρχει ανάγκη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά χωρίς να περνάμε από τη διαδικασία Άμπλετ ή πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει βελτίωση της διαδικασίας αυτής ώστε να καθισχαστούν οι ανησυχίες και βλέπετε πρόβλημα οι τρίτες χώρες οι οποίες βέβαια εφαρμόζουν αμοιβαιότητα στο διεθνές δίκαιο και άρα έχουν και αυτές πρόσβαση στα δεδομένα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και άρα στα δεδομένα των Ευρωπαίων με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υπάρχει πρόσβαση αυτή και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριε Σίπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω γερμανικά. Ζητώ συγγνώμη, δεν παρακολούθησα όλη την ε, ομιλία. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να συζητήσω με αστυνομικού στη Γερμανία, όπου ένα πρόβλημα ήταν ότι η τεχνολογική εμπειρία για την δίωξη, η παρακολούθηση του τι συμβαίνει στο διαδίκτυο, το ανοιχτό ή το σκοτεινό, δεν υπάρχει. Υπάρχει απαραίτητη τεχνογνωσία ή τεχνικές δυνατότητες ε, για να παρέμβουν. Δεν θέλω να ξέρω τι γίνεται στην Europol, αλλά οπωσδήποτε έχει και κάποια σχέση με τις δομές της Εθνικές Αστυνομικές Αρχές ε, και με τα έσοδα. Ε, Θεωρείτε ότι έχουν αναγνωρίσει το θέμα αυτό τα κράτη-μέλη και μπορείτε εσείς να τους βοηθήσετε να το αναγνωρίσουν και να δουν πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Το δεύτερο είναι το ερώτημα πόσα άτομα θα χρειαζόταν για μια παρέμβαση στο σκοτεινό δίκτυο. Αν έχουμε κάποιο έγκλημα στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν ας πούμε κάποιοι οι οποίοι πηγαίνουν ως ε, μυστικοί αστυνομικοί. Ε, γίνεται κάτι τέτοιο γίνεται στα κρατημέλη. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με το grooming, ε, με το οποίο προσεγγίζουν οι παιδεραστές ε, τους ανήλικους. Ε, κάνετε κάτι για να ανακαλύψετε αυτούς τους ανθρώπους και να κάνετε κάτι μετά. Το άλλο επίσης πολύ προβληματικό ε, αφορά το πώς θα μπορέσουμε να εμποδίσουμε να ανεβαίνουν εξ αρχής τα εγκληματικά περιεχόμενα ή να κατεβαίνουν μετά. Ε, πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε κάποιον ο οποίος ανέβασε έναν αλγορίθμο τέλει, χωρίς ε, καμία αιτία και μετά ε, τον κατέβασε. Πώς βλέπετε τα πράγματα και ποιο είναι το όριο που θα πρέπει να παρεμβαίνουν οι ιδιοκτικές αρχές για να κρίνουν τι είναι νόμο και τι παράνομο. Τέλος για την κρυπτογράφηση είναι θα πρέπει νομίζω και πολύ περισσότεροι να λάβουμε υπόψη ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν την κρυπτογράφηση για να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους ε, από ότι εγκληματίε. Θα πρέπει να βρεθεί λοιπόν ένας έξυπνος ε, τρόπος ε, που δεν θα θέτει σε κίνδυνο την προστασία των δεδομένων. Ευχαριστώ κυρία Ζίπελ. Κυρία Μαν. κυρία Μαν. Έχετε τον λόγο. Well, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, ερωτήσεις σας. Ε, θα ήθελα βέβαια και να ευχαριστώ και την Επιτροπή Λίμπη για την υποστήριξη προς τη δουλειά μας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις όσο καλύτερα μπορώ. Ε, βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες ερωτήσεις δεν μπορώ να απαντήσω. Κυρία Ζήπελ, ξεκινάω με εσάς. Λοιπόν, για την κρυπτογράφηση. Πράγματι είναι πρόκληση για μας, αλλά μίλησα για την πρόληψη. Η κρυπτογράφηση είναι ακρογνέως ε, λίθος ε, των κυβερνοεγκλημάτων. Το 2016 μαζί με την ΕΝΙΖΑ είπαμε ότι δεν στηρίζουμε μέτρα που να αφορούν γενικά στην κρυπτογράφηση. το να χρησιμοποιούμε πίσω πόρτες, αυτό δεν θα το κάνουμε. Εμείς θέλουμε να στηρίζουμε νόμιμα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τη νόμιμη χρήση κρυπτογράφησης. Στηρίζουμε την εργασία των εμπειρογνωμόνων. Θα υπάρξει μια ολόκληρη σειρά μέτρων. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει τα μέτρα που θα ληφθούν να είναι ανάλογα ε, και νόμιμα, νομότυπα. Ερώτηση του κυρίου Στίβενς σχετικά με το περιεχόμενο του διαδικτύου σε σχέση με ε, κηρύγματα μίσους ή ε, τρομοκρατία. Υπάρχει μια μονάδα που ασχολείται με αυτά και νομίζω ότι αναπόκειται σε εμά να αποφασίσουμε επί του θέματος να μας πούν τα κράτη-μέλη τι ακριβώς επιθυμούν. Γνωρίζουμε τις συζητήσεις που διεξάγονται. Υπάρχει μια προσέγγιση που λέει ότι να προβάλλονται αντίλογοι αντί να αφαιρείται το περιεχόμενο. Η άλλη ερώτηση ήταν πόσοι χρειάζονται για να ε, ασχολούν και να ερευνούν το σκοτεινό δίκτυο. Χρειαζόμαστε πόρους, περισσότερους πόρους, ανθρώπινους πόρους. Ανθρώπους με δεξιότητες ε, και τεχνογνωσία, αλλά και οικονομικούς πόρους για να αγοράσουμε τα εργαλεία, τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος και πάλι το βασικό είναι ότι στηρίζουμε τα κράτη-μέλη. Όπως ξέρετε, εμείς δεν είμαστε ευρωπαϊκό FBI, είμαστε εδώ για να στηρίζουμε τις έρευνες στα κράτη-μέλη και στο βαθμό του δυνατού προσφέρουμε υπηρεσίες και σε αυτό, στα κράτη-μέλη. Είναι βέβαια λίγο πιο δύσκολο να αποκτήσει κανείς ε, ανθρώπινους πόρους αλλά και εργαλεία και εξοπλισμό. Και αυτό αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη προσφέροντας ε, κεντρικές υπηρεσίες, να μην δηλαδή προκύπτουν καταστάσεις όπου επαναλαμβάνεται τα ίδια και τα ίδια ε, και τεχνογνωσία, ε, η ίδια τεχνογνωσία στα κράτη-μέλη. Στόχος μας είναι να προβάλλουμε όλα αυτά τα θέματα Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν τις προκλήσεις που υπάρχουν σχετικά με το κυβερνοέγκλημα και το σκοτεινό δίκτυο. Και τι ακριβώς χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν αυτά αποτελεσματικά. Ένα βασικό μήνυμα είναι ότι καμία υπηρεσία, αλλά δηλαδή και κανένα κράτος μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ε, τα θέματα αυτά, γιατί πλέον δεν έχουν σύνορα, είναι διεθνή. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους. Εμείς ως ε, Europol κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίζουμε τις έρευνες των κρατών μελών, να συγκεντρώνουμε σε κεντρικό σημείο την τεχνογνωσία. Ευχαριστώ και τους ε, άλλους ομιλητές και τους ευρωβουλευτές για όλα αυτά που είπαν. Ε, πράγματι υπάρχουν νομικές ε, προκλήσεις για να αντιμετωπιστούν τα διάφορα στοιχεία που προκύπτουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής. Ε, δεν είμαι και δικηγόρος, δεν μπορώ νομικά να σας απαντήσω ε, τι θα έπρεπε να κάνουμε ε, για να ξεκινήσει μια σχετική διαδικασία. Αν δούμε το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιταχύνει τη διαδικασία αυτό ήδη ε, είναι κάτι σημαντικό και υπάρχουν και άλλοι που συνεργάζονται πάνω σε αυτό νομίζω ότι ε, μπορούμε τη διαδικασία να την κάνουμε πιο αποτελεσματική και αυτό που έχει σημασία είναι ότι όποια διαδικασία και αν διαλέξουμε αυτή θα πρέπει να είναι νομότυπη, ανάλογη και απαραίτητη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αλλά σας είπα από πλευράς νομικής ε, δεν μπορώ να σχολιάσω, δεν μπορώ να μπω σε νομικές ε, λεπτομέρειες. Και σχετικά με αυτό πρώτος ο κύριος Στίβενς, ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας, ε, αλλά να ξαναπώ ότι υπάρχουν τεχνικές λύσεις για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε παράνομο περιεχόμενο ή κάποιες μορφές περιεχομένου στο διαδίκτυο. Τώρα, το πώς όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται και με ποιο τρόπο πρέπει να αντιδρούμε και πάλι δεν εναπόκειται σε εμά να αποφασίζουμε αλλά ε, στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας και για την παρουσία σας εδώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη τώρα. και θα ακούσουμε για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το Eurojust. Ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων. 19 Οκτωβρίου ε, το συζητήσαμε στην Επιτροπή μας, ξεκίνησε ο τριμερής διάλογος, ο κύριος Φως η να δώσω σε εσάς το λόγο να περιμένουμε. Εσείς, η σειρά σα είναι. Κύριε Φω. Ενημερώστε μας παρακαλώ για τις διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσω Από τις αρχές του Νοεμβρίου υπήρξαν δύο γύρια διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και υπήρξε και μία μικρή διάρκεια συνάντηση με τους και ηγητές. Ε, εστιάσαμε λοιπόν την προσοχή μας σε τέσσερις τεχνικές ε, συναντήσεις και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει και άλλη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών και εκεί ε, θα συζητήσουμε διεξοδικά για τα αποτελέσματα που εντωμεταξύ θα έχουμε επιτύχει και θα υπάρξουν και προετοιμασίες για την επόμενη συνεδρίαση. παρότι λοιπόν δεν με πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, σημειώσαμε ικανοποιητική πρόοδο σε πολιτικό επίπεδο, ε, εξετάσαμε τα θέματα, τα άρθρα, με συγχωρείτε, 1 έως 20, επεξεργαστήκαμε και αρκετές συμβαστικές προτάσεις. Υπάρχουν όμως κάποια ε, προσκόμματα, εκεί δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε. Αφενός το άρθρο 3, παράγραφος 1, ε, το οποίο αφορά την κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στη Eurojust και τον Ευρωπαίο εισαγγελίων ε, έχουμε ήδη διασφαλίσει το πρώτο σχέδιο συμβιβασμού. Θα το λάβουν υπόψη στα κράτη-μέλη, κυρίως εκείνα που δεν θέλουν να συμμετέχουν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Όμως υπάρχουν και άλλα θέματα που παραμένουν αντιευκρίνιστα Υπάρχουν και κάποιες ε, ε, αξιόπινες πράξεις που απαριθμούνται, ε, οι οποίες πράξεις όμως αυτές εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Eurojust. Δεύτερο επίμαχο θέμα, το 3, άρθρο 3, παράγραφος 4. Το θέμα είναι κατά πόσον οι έρευνες τις οποίες διεξάγει η Eurojust μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά πόσον οι έρευνες αυτές θα εξαρτώνται από τη συγκατάθεση ενός κράτους μέλους. Επ' αυτού δίστανται οι απόψεις. Βεβαίως το Συμβούλιο πιστεύει ότι το αρμόδιο κράτος το κράτος που, αφο, που εμπλέκεται θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του. Και θα δούμε με άλλες τεχνικές συζητήσεις που θα ακολουθήσουν θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Κατά τη δική μας την άποψη ισχύει το εξής. Ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει έτοιμα προς τη Eurojust, αυτό δεν σημαίνει ότι το, εμπλεκόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα της αρνησικυρίας. κυρίας. Ε, δεν θα πρέπει να μπορεί να ε, σταματά τις έρευνες. Στα άρθρα 10 και 11 που αφορούν ε, στην σύνθεση του κολεγίου, όπως επίσης ε, και το αξίωμα του Πρόεδρου και του Αντιπρόεδρου και από αυτό υπήρξε κάποια διάσταση απόψεων. Παραδείγματο χάρη ε, θα υπάρξει συμβασμο για το θέμα της εκλεγής ε, του Πρόεδρου. Βέβαια το Συμβούλιο εξακολουθεί να κάνει λόγο για κάποιο μηχανισμό αποζημίωσης γιατί κατ' ουσίαν το αξίωμα του Πρόεδρου για μικρά κράτη-μέλη θα συνεπάγεται υψηλέ δαπάνε. Άρα αυτά τα κράτη θα πρέπει κάπως να αποζημιώνονται. Πάντως ε, ε, κάπως πλησιάζουμε προς το θέμα αυτό, προς το να βρεθεί μια λύση ε, και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την εντύπωση ότι ε, άλλη λύση καλύτερα να βρεθούμε από το να προβλέψουμε άλλη μία αποζημίωση. Στα άρθρα 5 και άρθρο 14 εκεί έγινε συζήτηση για τις ενέργειες διαχείρισης ε, του κολεγίου και ε, όλοι συμφώνησαν, συμφώνησαν ότι ε, το διοικητικό φορτίο θα πρέπει επ' αυτού να υπάρξει μια διεξοδικότερη συζήτηση και δεν συμφωνήσαμε επ' αυτού. Αν θέλετε, αυτά ήταν γενικά τα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν στη συζήτηση. Κατά τα άλλα, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, εκεί η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική διότι προκύπτουν ιδιαίτερα επίμαχα θέματα επειδή υπάρχει σχέση με την έκθεση Κονίλια Ernst προστασία δεδομένων για τους ε, θεσμούς και υπάρχουν ε, τελείως διαφορετικές απόψεις ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει σχετική πρόταση. Το Συμβούλιο επιθυμεί στο 45-2001 σε αυτό το πλαίσιο να μην συμπεριληφθεί απαραίτητα κάτι που να αφορά τις διοκτικές αρχές. Το Κοινοβούλιο όμως θέλει ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσουν οι, εκθε... συζητήσεις σε αυτή την έκθεση στο 45201 και μετά θα πρέπει και εμείς να αποφασίσουμε κατά πόσον θέλουμε για τη Eurojust ένα ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας δεδομένων ή να κάνουμε περίπου αυτό που κάναμε και στη Europol, δηλαδή διασύνδεση αυτού που λείπει στο 45-2001 και αυτού που ε, ενδεχομένως λείπει στη Eurojust. Παραλαμβάνω όμως όλα αυτά είναι ασαφή και εξαρτώνται από τον ε, τριμερή διάλογο για το 45-2001. Και θέλω να σας πω ότι τόσο η Europol όσο και το περίφημο Joint Supervisory Board ε, μας έστειλαν επιστολές και μας επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό για όλα αυτά να υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Όμως, εγώ θέλω να πω ότι βασικά ε, τώρα είμαστε ε, μέσα στον τριμερή διάλογο και να περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τον 45-2001. Υπάρχουν βέβαια οι δύο επιστολές που μας εστάλησαν και παραλάβαμε και οι επιστολές αυτές περιγράφουν την κατάσταση. Όλοι μας βέβαια θεωρούμε ότι ανεξάρτητα με το σε ποια λύση τελικά θα καταλήξουμε δεν πρέπει να υπάρξουν ούτε παρερμηνείς ούτε διαφορετικές ερμηνείες δύο διαφορετικών νομικών πράξεων και που δεν, είναι, δεν πρέπει όλα αυτά να είναι εις βάρος της ποιότητας και της πραγματικής εργασίας. Στον τριμερή διάλογο θα μεριμνήσουμε έτσι ώστε η Eurojust, γιατί μόνο στη Eurojust δεν μπορώ να αναφερθώ, η Eurojust να έχει συγκεκριμένες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, αυτές οι διατάξεις να καθορίζουν την εργασία της και να συνεχιστεί η εργασία της Eurojust ακριβώς στο ίδιο ικανοποιητικό επίπεδο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Επιτροπής, της Εστονικής Προεδρίας, της Γραμματείας της Επιτροπής μας, αλλά και τους σκιώδης ηγητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγαστή συνεργασία. Καλό κλίμα επικράτησε ανάμεσα σε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Και γι' αυτό το λόγο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατορθώσουμε να επιτύχουμε τόσα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βόσου. Ποιο θέλει να πάρει το λόγο. Κανείς, τότε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε να προσθέσετε κάτι. Ναι. Σύντομα παρακαλώ. Θέλω να συμφωνήσω όμως, είπε ο κύριος Βός. Η καλή ατμόσφαιρα έχει να κάνει με το δικό του αισθητήριο χιούμορ, το οποίο πολύ βοηθάει. Και έτσι μας κάνει να νιώθουμε όλοι πιο άνετα. Και έτσι προχωρούμε σε καλές συμφωνίες για όλα τα σημεία, συμβιβασμούς. Εκεί που πράγματι βλέπω πρόβλημα είναι στο καθεστώς συλλογής δεδομένων. Πράγματι πρέπει να δούμε εκεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των άλλων τριμερών διαλόγων για το 45-2001. Ελπίζω ότι θα υπάρχει ικανοποιητική λύση τελικά για όλους και ότι ο οργανισμός αυτός θα διέπεται από σαφήνεια και ότι οι εποπτικές εκθέσεις για τους δύο οργανισμούς ε, είναι κάτι που το θέλουν. Και αφού το θέλουν πρέπει να τους το δώσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί πάντως μέσω μιας διτής προσέγγισης. Να υπάρχει το γενικό καθεστώς του 45-2001 με το νέο κεφάλαιο 8α που προσθέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνούμε με την προσέγγιση αυτή. Και από εκεί και πέρα να υπάρχουν ε, ιδιαίτεροι κανόνες για τις περιπτώσεις που αφορούν τον ένα τον άλλον οργανισμό και τη νομική του βάση. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε γρήγορα να προχωρήσουμε σε ένα συμβαστικό κείμενο για τα σημεία τα οποία απομένουν, όπως είπε και ο κύριος Φως. Και ελπίζω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα το έχουμε καταφέρει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρος. Κύριε Τσόνκα και εσάς κύριε Φως. Και τώρα... Είναι νωρίτερα από την ώρα μας, αλλά να ρωτήσω την κύριε Τίγκαν, είσαστε έτοιμοι να μας παρουσιάσετε την έκθεση προόδου που είναι το τελευταίο μας ε, σημείο για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση και την πέμπτη έκθεση για την άνοιξη υπηρεσιακής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Συναριοφυλακής και Εκτοφυλακής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας κάνει αυτή την παρουσίαση και θα μας μιλήσει και για τις εφαρμοστικές εκθέσεις και για την μετεγκατάσταση και για τη συμφωνία με την Τουρκία και για την κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Η ε, κυρία Τσιγκάν λοιπόν που είναι διευθύντρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει αυτό το θέμα που σίγουρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παρακαλώ κύριε Τσιγκάν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω με τον το θέσω στο γνωστό πλαίσιο από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη μετανάστευση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της μεταναστευτικής πολιτικής. Έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση και στην ανακοίνωση που παρουσιάσαμε και στην Επιτροπή σας, στην ανακοίνωση της ε, Κομισιόν. Παρουσιάσαμε την ε, γενικότερη αξιολόγηση του προγράμματος αυτού, την εφαρμογή του και όσον αφορά την αντίδραση στην κρίση και στις εξελίξεις αυτής της ε, τσάντας. Και ένα από τα μέσα για να μετρήσουμε την πρόοδο και να δούμε το πού βρισκόμαστε στην εφαρμογή είναι οι τακτικές εκθέσεις. Μέχρι στιγμής αυτό γίνεται με τρόπο κατακαιρματισμένο. Συντάσσουμε εκθέσεις που αφορούν συγκεκριμένα θέματα που είναι τμήματα της Ευρωπαϊκής Ατζέντα για τη Μετανάστευση, αλλά στις 15 Οκτωβρίου προτείναμε την πρώτη ενοποιημένη έκθεση πρόοδου που περιλαμβάνει όλα τα τμήματα τα οποία αφορούσαν ακριβώς ε, τα ζητήματα αυτά, την δήλωση με την Τουρκία, η εφαρμογή στα θέματα με την κατάσταση, επιχειρησιακή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και πλαίσιο συνεργασίας. Νομίζω ότι βοηθάει πολύ να έχουμε ένα συνολικό πλαίσιο της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε το τι γίνεται στην πράξη επιτόπου και θα μας βοηθήσει εν ώψη των επόμενων βημάτων. Εδώ πέρα δηλαδή το Δεκέμβριο θα έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οπότε έχουμε ένα πάρα πολύ καλό έγγραφο που περιέχει πολλές πληροφορίες που θα διαβιβαστεί σε όλους με τρόπο διαφανή. Η έκθεση ξεκινάει και θα ξεκινάει με την παρουσίαση της ε, κατάστασης που βασίζεται στα δεδομένα μας εδώ πέρα έχουμε όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε για να δείξουμε πώς έχει η τρέχουσα κατάσταση σε διαφορετικά σημεία. Βλέπουμε λοιπόν από την έκθεση πως η κατάσταση είναι η εξής. Οι κινήσεις είναι περιορισμένες στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο αριθμός ανείχνευσης ε, παρατύπων μεταναστών έχει σταθεροποιηθεί σε ένα χαμηλό επίπεδο στα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, η κεντρική Μεσόγειος εξακολουθεί να, είναι, να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, αν και με μια τάση μειούμενη από τα μέσα Ιουλίου και μια ανωδική τάση καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του 2017 στην Δυτική ε, Μεσόγειο και Ατλαντικό. Θα ξεκινήσω τώρα με κάποιες πληροφορίες που αφορούν τα διάφορα τμήματα, αλλά αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Θα ξεκινήσω προφανώς με την επιχειρηματική επιχειρησιακή ή ικανότητα για να αντιδράσουμε σε μια κατάσταση κρίσης. Πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε εδώ τα hotspots στην Ελλάδα και την Ιταλία ότι αξιολογήσαμε την λειτουργία τους μέχρι στιγμής και είδαμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, όσον αφορά την προσέγγιση μας και είδαμε συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να βοηθηθούν τα παιδιά και ευπαθείς ομάδες και όπως έχουμε πει επανειλημμένως εδώ στην Επιτροπή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για την έννοια του hotspot δηλαδή δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει μια καλή επιχειρησιακή συνεργασία των υπηρεσιών μας τώρα για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές πληροφορίες στην έκθεση αλλά η τρέχουσα προτεραιότητα είναι η μεταφορά όσο δυνατόν περισσότερων από τα στρατόπεδα σε νοικιαζόμενη στέγη καθώς ε, οι ελλείψεις ε, του συστήματος ε, είναι επίμονες. Γνωρίζω πως είχατε μία αναλυτική παρουσίαση της προετοιμασίας για τον χειμώνα και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τον Επίτροπο τον κύριο Αβραμόπουλο στην Ολομέλεια για την εφαρμογή της δήλωσης με την Τουρκία έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα στην μείωση παρατύπων δύο άδελων και σώζονται έτσι ζωές. Όμως οι επιστροφές στην Τουρκία είναι πολύ χαμηλές. Η επανεγκατάσταση από την Τουρκία συνεχίζεται και βεβαίω πρέπει να διατηρηθεί ο ψηλός ρυθμός. Συνολικά από τον Απρίλιο του 2016 πάνω από 14.000 άτομα έχουν μετεγκατασταθεί από την Τουρκία. Νομίζω επίσης πως πρέπει να αναφέρουμε εδώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε καλό δρόμο για να διαθέσει τα 3 δισεκατομμύρια στο μέσο των προσφύγων στην Τουρκία μέχρι το τέλος του έτους. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι οι πληροφορίες για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν πίεση μετά από την κρίση στη Συρία όπως ο Λίβανος και η Ορδανία Συνεχίζεται, αλλά είναι επίσης σαφές ότι υπάρχει ανάγκη διεθνούς οικονομικής στήριξης που θα πρέπει να συνεχιστεί και νομίζω πως ε, θα φανεί αυτό και το έχουμε βάλει ως ε, σημείο αναφοράς. Θα το δούμε λοιπόν στην διάσκεψη των Βρυξελών την ερχόμενη άνοιξη την διάσκεψη για την Συρία που θα συζητήσουμε. Τη της οικονομικής στήριξης. Για την Κεντρική Μεσόγειο έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι. Περιγράφει την επιχειρησιακή μας αντίδραση, το μεγαλύτερο κομμάτι δράσης που αφορούν την Λιβύη. Η έκθεσή μας αναγνωρίζει, διαβάζω, τι συχνά αποκρουστικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μεταναστές στη Λιβύη, τα γνωρίζουμε, αλλά τονίζει την σύγχρονη έπαφη μας και δέσμευσή μας για να βελτιωθεί η κατάσταση στο πλαίσιο αυτό. Θα ήθελα να φέρω ιδιαίτερα τις ε, δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση της ε, Λιβικής Ακτοφυλακής, το πρόγραμμα 90 εκατομμυρίων για να βελτιωθούν οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν στη Λιβύη οι μετανάστες και βεβαίως ε, σχετίζονται εδώ πέρα και οι διαφορές δράσεις υποδομής, έχουμε το συγκεκριμένο κομμάτι που αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα και υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες που αφορούν την χρήση του ταμείου και βεβαίω τα των επενδύσεων και των υπεργολαβίων και το ποιο είναι το κενό το χρηματοδοτικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με την Πατερμοστία του και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για τις εθελοντικές επιστροφές και την επανένταξη ε, στην διαδρομή της κεντρικής μεσαγίου και στα σημεία αποβίβασης και στα κέντρα κράτησης. Μία σύντομη αναφορά στα άλλα σημεία. Η έκθεση επιβεβαιώνει πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για να σταματήσει το επιχειρηματικό μοντέλο των ε, διακινητών. Στο πλαίσιο αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες ε, μεταξύ κρατών μελών, αποστολών ΚΕΠΑ και να επεκτείνουμε τις ε, κοινέ ομάδες έρευνων με χώρες Δυτικής Αφρικής. Νομίζω πως στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να ενημερώσουμε για όλες αυτές τις δραστηριότητες στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στα κράτη-μέλη τους πολίτες μας νομίζω ότι πολύ συχνά δεν γνωρίζουν τα αποτελέσματα και ότι υπάρχουν και ουσιαστικά αποτελέσματα στα κράτη-μέλη και νομίζω πως έχει σημασία να γίνει αυτό γιατί το ε, σπάστο το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών είναι νομίζω το σημαντικότερο. Τώρα, για τις επιστροφές και την επανεισδοχή νομίζω πως είχατε συζητήσεις, ε, ναι, είχατε εδώ πέρα και τον ε, υποδιευθυντή μας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα αναφερθώ σε δύο στοιχεία που είναι στην έκθεση προόδου. Αναφερόμαστε εκεί στην ανάγκη να υπάρχουν έγκαιρα και έγκυρα δεδομένα για τις επιστροφές. Δεν είναι μόνο ζήτημα αριθμών, αλλά υπάρχει μια καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης έτσι. Και εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα εσωτερικά, αλλά συνεργαζόμαστε και με την Eurostat για να έχουμε αυτά τα δεδομένα και να τα συλλέγουμε πιο συχνά και με καλύτερο τρόπο και θα αναφερθώ και στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Νοέμβριο το οποίο αφορούσε τα έπιχησιακά βήματα για να αρχίσουν οι επιστροφές και ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να επενδύσουν περισσότερο στο προσωπικό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια δέσμευση για να υπάρξει ένα πλαίσιο επιστροφών. Θα πω τώρα λίγα λόγια για την υπηρεσία αυτή. Στο τέλος της ομιλίας μου για, τις, ε, ε, ε, για τους υπηρεσίες EBCGA και ECGA. Όσον αφορά την επανεγκατάσταση και τη μετεγκατάσταση, οι συζητήσεις έχουν γίνει με λεπτομέρειες εδώ στην Επιτροπή. Γνωρίζετε ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τη μετεγκατάσταση. Πάνω από 31.000 άνθρωποι έχουν μετεγκατασταθεί και αυτό δείχνει ότι ε, και μετά τις 26 Σεπτεμβρίου εξακολουθούμε να στηρίζουμε την ε, μετεγκατάσταση. Ε, 140 ετούντες ε, δεν έχουν ακόμα μετεγκατσαθεί από την Ελλάδα και περίπου 200 από την Ιταλία. Υπάρχουν ε, κάποιες δράσεις ε, που πρέπει να ολοκληρωθούν για να ολοκληρωθούν και τα σημαντικότερα βήματα. Ε, τα αναφέρω αυτά και στην έκθεση πρόοδου. Ε, αναφέρω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ε, δικαιούχοι νομότυποι μετανάστες για μετεγκατάσταση Ενημερώνω επίσης και για επιπρόσθετες θέσεις που μπορούν να προσφερθούν κυρίως για συνόδευτα ε, παιδιά από την Ιταλία. Και τέλος ε, γίνεται λόγος ε, και για τις υποσχέσεις, για όλα αυτά που δεν έχουν ακόμα λάβει χώρα. Όσον αφορά την την επαναγκατάσταση. 22.000 ήταν το 2015, 81% έχει ε, ολοκληρωθεί, 80.000 ε, έχουν επαναγκασταθεί σε 28 κρατημέλη μελη Οι περισσότεροι ήρθαν από την Τουρκία, την Ιορδανία και το Λίβανο. Και μετά ε, την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη-μέλη να προσφέρουν τουλάχιστον άλλες 15.000 θέσεις επαναγκατάστασης. Μέχρι τώρα 17 κρατημέλη έχουν δεχτεί πάνω από 34.500 προσφέρουν δηλαδή αυτές τις θέσεις επαναγκατάστασης και ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλες υποσχέσεις για να επιτευχθεί ο στόχος. Θα ήθελα να αναφέρω και κάποιες πληροφορίες για πιλωτικά προγράμματα που αφορούν στην ομότυπη μετανάστευση. Αυτά ήδη ανακοίνονται στην ανακοίνωση της 27ης Σεπτεμβρίου. Προτείνουμε πιλωτικό πρόγραμμα για την νομότυπη μετανάστευση ε, στα κράτη-μέλη που δέχονται ε, κάποιους μετανάστες. Εμείς ε, προτείνουμε και να στηρίξουμε την ενσωμάτωση των μεταναστών σε όλες τις φάσεις προετοιμασία ε, της νομότυπης μετανάστευσης και μετά την ενσωμάτωση των μεταναστών σε διάφορους ε, τομείς. Επίσης ε, θα συνεχίσουμε να συζητάμε με τα κράτη-μέλη για προγράμματα και υποψήφιους μετανάστες. Ε, οι συνθήκες αναφέρονται σε αυτή την ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου. Εκεί γίνεται αξιολόγηση και της ε, λογικής ε, πίσω από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Αυτά είχα να πω για την έκθεση προόδου της 15ης Νοεμβρίου. Ε, όσον αφορά το EBCG, ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία σε αυτή την έκθεση της 15ης Νοεμβρίου, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα ε, στην έκθεση που είχε εγκριθεί νωρίτερα στις 6 Νοεμβρίου. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε αυτά τα στοιχεία. Νομίζω όμως ότι ε, είναι πολύ καλή ευκαιρία που προσφέρεται σήμερα γιατί έχουμε και το παράρτημα της τελευταίας έκθεσης ε, πρόοδου ε, που περιλαμβάνει επιπρόσθετες πληροφορίες σε αυτές που παρουσιάστηκαν το Σεπτέμβρη. Είναι επίκαιρε οι πληροφορίες και στην περίπτωση αυτή θέλω να πω θα θυμάστε όλοι την το νομοθετικό πλαίσιο για αυτό τον φορέα BCG χρειαστήκαμε νέα μήνες και τώρα πλέον είμαστε εννέα μήνες μετά την ε, εφαρμογή αυτού του πλαισίου. Ε, πλέον ε, νομίζω ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ουσιαστικά. Πρέπει να αναφέρουμε τα επιτεύγματα και όπως το κάνει και η έκθεση, να αναφέρουμε και κάποιες τομείς όπου είναι απαραίτητο να υπάρξουν βελτιώσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι ο φορέας ήδη προσφέρει ε, υποστήριξη στα κράτη-μέλη στη διαχείριση των ε, συνόρων, ε, περίπου 1500 παραμεθόροι φρουροί έχουν προσφερθεί Χρειάζονται βέβαια περισσότερες προσπάθειες. Δεν πρόκειται μόνο για τον αριθμό του προσωπικού αλλά και για τους εμπειρογνώμονες που είναι απαραίτητοι. Χρειάζονται λοιπόν ε, συγκεκριμένες διευκρινήσεις ε, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή EBCG. Αυτά λοιπόν πρέπει να βελτιωθούν. Η έκθεση προόδου ε, έχει κατατεθεί, αλλά εντωμεταξύ υπάρχουν και επικαιροποιήσεις κάθε εβδομάδα. Αυτό βοηθάει ε, στο να καλούμε τα κράτη-μέλη να κλείσουν τα χάσματα που υφίστανται. Σχετικά με την μονάδα ε, ταχείας αντίδρασης και τη σχετική δεξαμενή που πρέπει να σχηματίσουμε υπάρχουν κενά γιατί μέχρι τώρα έχουν συμβάλει μόνο 14 κράτη-μέλη. Σας είπα ότι έχουμε πάνω από 1.500 ε, σύνοριοφύλακες, 26 ε, κράτη-μέλη έχουν ορίσει αυτούς τους ε, σύνοριοφύλακες, άρα δηλαδή το 74%. Το δεύτερο που θέλω να, βέλω, να αναφέρω είναι το στοιχείο του, των αξιολογήσεων περί του ευάλωτου στοιχείου της αδυναμίας που μπορεί να εφίσταται. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένες ε, προτάσεις ε, σχετικά με αποτελεσματικό έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς αυτή τη διαδικασία τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Γιατί λαμβάνουμε υπόψη μας ότι Υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν προκύψει από την αξιολόγηση της Συμφωνίας Σέγκεν και από άλλες μελέτες για καλύτερη χρήση των πόρων. Ένα άλλο που θέλω να φέρω αφορά τη διεθνή συνεργασία. Εδώ έχουν γίνει συζητήσεις ε, με την ΦΥΡΟΜ, οι συζητήσεις αυτές συνεχίζονται τον Οκτώβρη το Συμβούλιο έδωσε πράσινο φως στην Επιτροπή να ε, διαπραγματευτεί παρεμφερή συμφωνίες με την Αλβανία, το Μαυροβούνι και τη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Επόμενο επίτευγμα είναι μια στρατηγική για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων. Αυτή η στρατηγική πρέπει ε, να χαράστε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εργασίες συνεχίζονται και εργαζόμεθα για την ε, προετοιμασία της ανακοίνωσης. Και τέλος, η συμφωνία σχετικά με την έδρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και την Ακτοφυλακή και την Πολωνία, ανάμεσα αυτούς τους δύο, ετέθη αρχές Νοεμβρίου ε, σε ισχύ αυτή η συμφωνία και προσπαθούμε να βρούμε τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την καλύτερη λειτουργία της ε, συνοριοφυλακής και εκτοφυλακής. Νομίζω ότι καταλάβατε ότι μπλεκόμεθα σε διάφορες φάσεις και σε διάφορα επίπεδα. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σα έχει ενημερώσει σχετικά με την αξιολόγηση του τι είναι τροτό, ποια είναι τα τροτά σημεία Είχαμε μία συνάντηση υψηλού επίπεδου ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη και αυτό είναι μία σημαντική πηγή πληροφοριών για μας. Πληροφορίες τις οποίες ε, θα εκμεταλλευτούμε για να χαράξουμε σωστή στρατηγική για τη σωστή διαχείριση των συνόρων. Και ολοκληρώνοντας ε, θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή παραμένει πρώτη προτεραιότητα για όλους μας και θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας. Αυτά είχα να σας πω εν είδη εισαγωγής και ευχαριστώ στη διάθεσή σας αν έχετε σχόλια και ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σιγκάλ για την τόσο πλήρη παρουσίασή σας. Οι συνάδελφοι τώρα. Ποιος θέλει το λόγο η κυρία Κέλλερ, η κυρία Βερζιά. Ωραία. Η κυρία Σίπελ μετά. Η κυρία Κέλλερ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την ε, παρουσία. Έχασα τα πρώτα λεπτά, αλλά νομίζω ότι το κυρίως μήνυμα το πήρα. Έχω κάποιες ερωτήσεις, παρακαλώ, και κάποιες παρατηρήσεις. Για τη Λιβύη θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε και στην Ολομέλεια. Επίγει να το κάνουμε. Όπως όλοι ξέρουμε, η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Και να νομίζουμε ότι ενισχύουμε τη συνεργασία όταν δεν λύνουμε τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν δεν τα αντιμετωπίζουμε τέλο πάντων ή τέλο πάντων δεν τα αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν, ε, νομίζω ότι είναι πράγματι ανυπόφορο. για το θέμα της μετεγκατάστασης. Όντως δεν έχουν γίνει οι προσπάθειες που θα έπρεπε να γίνουν από τις χώρες μέλη. Ελπίζω να συνεχίσει και η Επιτροπή να πιέζει τις χώρες μέλη. Και έχω μια ερώτηση για τη Frontex. Είπατε 74% του δυναμικού της ακτοφυλακής, έτσι είπατε. Και όταν ετοιμάσαμε την έντολη είχαμε προβλέψει κυρώσεις για όποια χώρα δεν τηρεί τις συστάσεις της Frontex όταν θα γινόταν κλείσιμο συνόρων ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είδαμε όμως τίποτα τέτοιο όταν μια χώρα δεν φροντίζει με πλήρη ποσόστοση να καλύπτει την ακτοφυλακή. Οπότε δεν μπορεί όλες οι χώρες να τα βάζουν με μία χώρα επειδή δεν κάνει αυτό που πρέπει, αλλά απ' την άλλη να είναι πρόθυμοι για κυρώσει. Λοιπόν, βασίζομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει τις χώρες μέλη ώστε 100% να τηρήσουν την ποσόστοσή τους. Θυμάμαι ότι είχαμε πει ότι έχουμε ένα πουλ με ξέρω εγώ πόσους ε, σε δυναμικό της ακτοφυλακής και τώρα μιλάμε για 74%. Και έχω και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Γίνονται πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα δικά μας εξωτερικά σύνορα και από τους δικούς μας. Δεν μιλάω για τη Frontex εδώ, από την εκτοφυλακή συνοριοφυλακή των χωρών μελών. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε άλλη μια περίπτωση, έξι χρονών ένα κοριτσάκι πέθανε στα συνορα κροατια Κροατίας-Σερβίας, γιατί είπανε στην οικογένεια να ακολουθήσει μια διαδρομή πίσω στη Σερβία η Κροατία τους είχε διώξει, δηλαδή πρέπει να πάνε πίσω στη Σερβία. Δεν βλέπανε το τρένο που ερχόταν, ήταν νύχτα και το παιδάκι πέθανε. γιατί τους είχαν βάλει να περπατάνε στη συνδρομική γραμμή. Ξέρω ότι η Επιτροπή θα πει χώρες μέλη φταίνε. Εντάξει, οι χώρες είναι υπεύθυνε, αλλά δεν είναι ικανοποιητικό να έχουμε από την άλλη μεριά μια Ευρωπαϊκή Ένωση με επιμερισμένη ευθύνη, με κοινά εξωτερικά σύνορα, με μια υπηρεσία υπεύθυνη γι' αυτό, να έχουμε κοινέ αξίε κτλ. και να μην είμαστε σε θέση να κάνουμε τίποτα για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βλέπουμε στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από συνοριοφύλακες μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μου πει τι σκέφτεται από αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτήν την πρώτη εκθεσή της, παρουσίασή της. Η πρώτη μου ερώτηση είναι ότι από τις 13 Μαρτίου 2015 τροποποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη μετανάστευση. Είχε τέσσερις προτεραιότητες τότε το Μάιο να μειωθεί η παράτυπη μετανάστευση, αυτό το πετύχαμε νομίζω, να σώσουμε ζωής και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στα σύνορα. Ε, για το δεύτερο, ναι, για το πρώτο δεν νομίζω. Τρίτον, να κάνουμε παραπάνω προσπάθειες για να πετύχουμε περισσότερο όσον αφορά το άσυλο, γιατί και εδώ έχω πάρα πολλέ αμφιβολίες. Ναι, κάποιες χώρες κάνουν παραπάνω προσπάθειε αλλά συνολικά όχι. Και τέλος, ναι, μεταναστευτική πολιτική για την επίσημη μετανάστευση. Αυτή η νόμιμη οδή που εμείς ζητούμε για την ε, νόμιμη μετανάστευση. Πούντι. Η επανεγκατάσταση δεν μπορεί να είναι η μόνη οδός. Αν υπήρχαν περισσότερες νόμιμοι οδοί για νόμιμη μετανάστευση από όλε αυτές τις χώρες, πρώτον θα είχαμε λιγότερη παράτυπη μετανάστευση και δεύτερον θα είχαμε και λιγότερους λαθρέμπορους, έτσι λιγότερους ε, λαθροδιακινητές. Τώρα θέλω να επικεντρωθώ στη Λιβύη. Φυσικά έχουμε επανέλθει στα επίπεδα του 2014, εντάξει. Σήμερα κοίταζα πάλι ένα παιδάκι τριών χρονών σώθηκε ως εκθαύματος από ένα πλοίο του SOS Μεσόγειος. Ακόμα και σήμερα δηλαδή άνθρωποι πνίγονται στη Μεσόγειο. Και αυτό που μας λένε όλο και περισσότερο οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και θα ήθελα η αλήθεια ε, να μην βγει όπως βγήκε στη Λιβύη. Μας λένε ότι υπάρχουν θάνατοι στην έρημο και ακόμα περισσότεροι σήμερα στην έρημο από ό,τι στη Μεσόγειο. Και εμείς τι κάνουμε, τους σπρώχνουμε πιο πολύ νότια, πιο πολύ στην έρημο. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό. Όταν πήγαμε στην Ισία, είχαμε όλε τις ε, πληροφορίες. Αυτά που μας είπε το CNN μετά δηλαδή, δεν ήταν έκπληξη για κανένα, τα ξέραμε. Όμω, όταν διαβάζω εδώ τις δύο παραγράφους στην έκθεση που είναι αφιερωμένε στη Λιβύη, ε, πραγματικά μένω με το στόμα ανοιχτό. Αυτά που λέει εδώ η έκθεση δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, στα όσα λέμε και ξαναλέμε για την κατάσταση στη Λιβύη πού πάνε τα χρήματα, σε ποιον πάνε τα χρήματα τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τι χρησιμεύουν. Μας λένε στις διεθνείς οργανώσεις. Ναι, αλλά κανένας δεν ελέγχει την επικράτεια της Λιβύης εκτός από τους παραστρατιωτικούς. Κανένας δεν έχει τον έλεγχο της επικράτειας. Οπότε τελικά πού πάνε τα χρήματα αυτά. Και όταν μας λένε ότι 2.000 οικογένειες βοηθήθηκαν, ότι 14 βοηθήθηκαν στα κέντρα, στους καταβλισμούς. Μα ποιος τους έλεγε τους καταβλισμούς αυτούς, οι παραστρατιωτικοί. Δεν ε, αλλάζει τίποτα εκεί επί της ουσίας. Να δούμε τα πράγματα όπως έχουν κατάματα. Εντάξει, θα γίνει η αποστολή αυτή αλλά πρέπει να ξέρουμε συγκεκριμένα σε ποιον δόθηκαν τα χρήματα αυτά, για ποιο λόγο και πώς χρησιμοποιήθηκαν. Γιατί πρόκειται για χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαίων, στους οποίους λογοδοτούμε. Δεν μπορεί να μας τάνουν αυτές οι δύο παράγραφοι. Για διαβάστε τες, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. δεν λένε τίποτα για όσα μας κατηγορούν. Και για το θέμα της μετεγκατάστασης, αν κατάλαβα καλά, η διαδικασία τελείωσε. Αν δεν υπάρξει νέα νομοθεσία, 169.000, τίποτα. Υπάρχουν 150 από την Ελλάδα και 300 από την Ιταλία που μετεγκαταστάθηκαν. Δεν υπάρχει δυνατότητα άλλη μετεγκατάσταση. Έτσι δεν είναι. Εκτό αν εμένα μου έχει ξεφύγει κάτι. Η επανεγκατάσταση μπορεί, αλλά όχι ή κατάσταση αν δεν υπάρξει νέα νομοθεσία. Και δεν το βλέπω να γίνεται σύντομα. Λοιπόν, είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Όχι, φοβάμαι. Υπενθυμίζω ότι η ατζέντα του Μαΐου του 2015 εγκρίθηκε πριν από την περίφημη κρίση ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα. Πριν. Μετά από ναυάγιο στα νότια της Λαπαντούσα όπου έχασαν τη ζωή τους 700 άνθρωποι σε μια μέρα. Τότε φτιάξαμε την ημερήσια διάταξη για τη μετανάστευση. Τώρα λοιπόν έχουμε επιστρέψει στα επίπεδα του 2014, πρέπει να έχουμε μια νέα ημερήσια διάταξη που να ανταποκρίνεται στα όσα εγκρίναμε το Μάιο του 2015. Ενώ είμαστε πολύ μακριά. Άκουσα να λέει η επιτροπή, α, τι κρίμα για τις επιστροφές στην Τουρκία. Ε, αυτό είναι ακρονάωτο μου φαίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας υπενθυμίσω ε, ότι αύριο το απόγευμα στις 2.30 θα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, κυρία Βερζιά, για την Λιβύη. Κυρία Τσίπελ. <laughs> Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε μόλις μία συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Πακέτο Ασύλου όπου παραπονεθήκαμε για το ότι η Κομισιόν, το Συμβούλιο, σε κάποια θέματα δεν έχει καν μια κοινή θέση. Τελείως διαφορετική είναι η κατάσταση στο θέμα της ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής. Το Συμβούλιο το ήθελε, κινήθηκε γρήγορα και τώρα έχουμε την πέμπτη έκθεση και ακόμα, αξόσον γνωρίζω, έχουμε μόλις 15 κράτη-μέλη που έχουν αποστείλει υλικό και προσωπικό ε, όπως ε, προβλεπόταν. Ε, λοιπόν, τι γίνεται. Πρώτα το θέλουν, το αποφασίζουν και μετά δεν κάνουν τα όσα υποσχέθηκαν ως παρατήρηση. Για να επανέλθω στην κατάσταση του μεταναστευτικού. Ε, τα λεφτά δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση και θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση εδώ για την Λιβύη. Ακούσαμε διαφορετικές οργανώσεις να μας λένε ότι αν δώσουμε λεφτά στη Λιβύη σε οποιονδήποτε τα άτομα αυτά, οι διοικήσεις, οτιδήποτε πρέπει να ε, δώσουν μέρος αυτών των χρημάτων σε συμμορίες αλλιώς δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Οπότε υπάρχουν και άλλα πράγματα εκεί και αντιλαμβάνομαι ότι η Κομισιόν, το Συμβούλιο, όποιο είναι, προσπαθεί να αναδιοργανώσει το κράτος στη Λιβύη. Αλλά ταυτόχρονα ακούμε συνεχώς για την καταστροφική κατάσταση για τους μετανάστες και κατά την απόψή μου είναι οδυνηρό να βλέπουμε ότι ο μόνος με μόνο στόχο να βρεθεί ένας τίτλος που θα λέει «Μειώνεται ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», θα δεχόμαστε την τραγική κατάσταση στη Λιβύη. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει μια σαφή διέξοδο από αυτή την κατάσταση. Και για τους Λίβιους που μπορεί να μην συμφωνούν με αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι είναι σε διαφορετική ε, φάση. Κάτι άλλο Μίλησα για τα λεφτά. Τι γίνεται με τα λεφτά για το Ταμείο για την Αφρική. Νομίζω ότι κάποια κρατημέλη δεν ε, δίνουν λεφτά. Πολλά από τα λεφτά προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Και τελευταία ερώτηση για τις διαδικασίες υπερβάσης βάρος κάποιων χωρών που δεν θέλουν να δεχτούν μια κατάσταση. Έχει να τίποτα νεότερο. Κύριε Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, εγώ ε, θα το αντιστρέψω λιγάκι. Θα ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, προσπάθειες που κατέβαλε, γιατί πιστεύω ότι και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη προχωράμε σιγά-σιγά. Ε, συνάδελφε, κατανοώ πλήρως αυτό που είπε σχετικά με, την, με το κοριτσάκι των έξι μηνών τώρα να μιλάμε για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιώματος ε, και δόλο. Δεν νομίζω ότι ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Θα έπρεπε να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί. Δηλαδή περισσότερο ήταν αμέλεια, ολιγορία και όχι δόλος. Πιστεύω ότι οι καταστάσεις ε, στα σύνορα ε, πολύ συχνά είναι πολύ πιο δύσκολες από αυτά που φανταζόμαστε εμείς στο Κοινοβούλιο και ε, δεν είναι έτσι απλό ότι ό,τι αφορά τους ε, πρόσφυγες να λέμε αυτά είναι καλά και ό,τι αφορά τους άλλους είναι δυσάριστα και αρνητικά. Ε, τα πράγματα είναι κάπου στη μέση, διαφοροποιημένα. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω για το ότι όλο και περισσότερα κράτη-μέλη όπως η Κροατία προσπαθούν να χειρίζονται καλύτερα το θέμα των προσφύγων. Έχουν αλλάξει θέση από αυτήν που είχαν πριν από 5-6 χρόνια. Συζητάνε πια και με τις συζητήσεις και με εμά σημειώνεται πρόοδος. Έχω κάποια ερώτηση προς την Κομισιόν σχετικά με το resettlement. Τα κράτη-μέλη εντωμεταξύ είναι έτοιμα να προχωρήσουν ε, περισσότερο από ό,τι κατά το παρελθόν σε σχέση με την μετεγκατάσταση ή εξακολουθούν να έχουν ε, έτσι κάποιες ε, διοικητικές επιφυλάξεις για να μην δέχονται πρόσφυγες στην επικράτειά τους είτε με μετεγκατάσταση είτε με επαναγκατάσταση. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλετε να απαντήσετε. Thank you very much and thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε και κύριοι βουλευτές για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω με μια σκέψη. Είναι σαφές ότι στην έκθεση πρόοδου και στην παρουσίασή μου αναφέρθηκα σε πολλούς αριθμούς. Δείτε όμως αυτούς τους αριθμούς, όπως είπα στην αρχή, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να δούμε το πώς έχει η κατάσταση, πώς εξελίσσεται η κατάσταση να έχουμε δεδομένα που θα μας δώσουν ολόκληρη την εικόνα και θα μας επιτρέψουν να δούμε κάποιες τάσεις. Με το να έχουμε λοιπόν τους αριθμούς που θα μας επιτρέψουν να προγραμματίσουμε καλύτερα και να γνωρίζουμε ε, δεν πρέπει βεβαίω να ξεχνάμε και τους ανθρώπους. Ε, δεν είναι δυνατόν. Ε, βεβαίως, το θέμα δεν είναι να ξεχνάμε τους ανθρώπους, είναι να έχουμε την δυνατότητα και τα μέσα να αξιολογήσουμε που, ε, πώς έχει κατάσταση. κάθε μετανάστης είναι άνθρωπος ε, και έτσι τους ε, εξετάζουμε. Κάθε απώλεια ζωής στη θάλασσα είναι τραγική και πάντα αυτή την αρχή ακολουθούμε. εντάξει, μπορώ να πω μόνο ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Αξιών. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι σημαντικά για εμάς. Έχουμε νομικές δεσμεύσεις που θα εφαρμόσουμε στις δράσεις μας. Προφανώς η κατάσταση είναι περίπλοκη. Αλλά σας διαβεβαιώ πως η συνεργασία μας με τρίτες χώρες η... ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ενσωματωμένος στα προγράμματα και βεβαίως ε, έχουμε και τους εταίρους από το σύστημα του ΟΗΕ και εκεί πέρα σε όλα αυτά ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό για μα. Παραδείγματο χάρη, μιλάμε για την Λιβύη και το τι μπορεί να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε για να ενισχυθεί ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και για την κατάσταση με την ε, Λιβική ακτοφυλακή. Αυτό είναι ένα κομμάτι και της εκπαίδευσης ε, που παρέχουμε και της διαδικασίας παρακολούθησης. Αν δούμε την κατάσταση του που πρέπει να πάνε τα λεφτά, κοιτάμε την κατάσταση των κέντρων κράτησης. Προσπαθούμε να υπάρξουν κάποιες τυποποιημένες ε, διαδικασίες στα μέρη αυτά. Στηρίζουμε τις δραστηριότητες, συνεργαζόμαστε με ανθρωπιστικούς οργανισμούς. Επίσης και στην πληροφόρηση των μεταναστών κάνουμε αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι μέρος της δουλειάς μας. Και όταν, αν δείτε το κομμάτι αυτό της έκθεσης πρόοδου για τη Λιβύη, είναι μια έκθεση πρόοδου. Το πλαίσιο της ανακοίνωσης του Σεπτεμβρίου, αλλά νομίζω ότι περιέχει μια ενδιαφέρουσα παράγραφο που αφορά τις υποδομές και το πώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις, ε, την οργάνωση της καθημερινής ζωής ε, των Λίβιων και των μεταναστών στηρίζοντας ε, μικρές επιχειρήσεις, την εκπαίδευση των παιδιών, βοηθώντας τις υφιστάμενες δομές και όπου υπάρχει χώρος για παιδιά και ενισχύοντας τις δυνατότητες της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Και λέμε ότι είναι δύσκολο το περιβάλλον στη Λιβύη και παραμένει μια πρόκληση, αλλά συνεργαζόμαστε ενεργά με τους εταίρους μας ε, που αναφέρονται για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους αυτούς. Οπότε η κατάσταση δεν είναι τέλεια, αλλά έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο για τη μετακατάσταση. Συμφωνώ απολύτως. Δεν επαρκεί και σας διαβεβαιώ ότι όλα τα μέτρα τα οποία λάβαμε απέναντι στα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή της αλληλεγγύης ε, συνεχίζουν. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία παραβάση και συνεχίζεται. την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και το 74% των ονομάτων. Ε, να διευκρινίσω κάτι γιατί μάλλον δεν εκφράστηκα σαφώς. Τα κράτη-μέλη επιβεβαίωσαν την διαθεσιμότητα των 1500 συνοριοφυλάκων και αυτή τη στιγμή οριστικοποιούν τα ονόματα. και μάλλον υπάρχει και μία καθυστέρηση γιατί υπάρχει βεβαίως ε, και το θέμα ακριβώς ε, των αποσπάσεων κτλ. Γιατί τα υπόλοιπα ονόματα πέρα από το 74% θα έρθουν όταν ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οπότε υποβάλλουμε τακτικές αναφορές και θα συνεχίσουμε και ελπίζω ότι με την περαιτέρω πληροφόρηση αυτή θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ολοκληρώσουν αυτήν την διαδικασία. Τώρα, για τις περιπτώσεις που γνωρίζετε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρακαλώ να μας κρατάτε ενήμερους. Ανέφερα συγκεκριμένα στην παρουσίασή μου το θέμα της ε, καταπολέμησης των διακινητών. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτό γιατί όλα τα παραδείγματα που μπορεί να δώσει κανείς ε, ξεκινάνε έτσι. Δηλαδή, ε, όσο αποτελεσματικοί και να γίνουμε, πάντα θα προσαρμόζονται. αν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι επίσης δεν έχουν έλεος και πάντα θα αντιμετωπίζουμε αυτές τις ε, καταστάσεις. Αλλά αυτός είναι ένας από τους πυλώνες της ε, δραστηριότητάς μας. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε πιο θετικά νέα προσεχώς. Και έτσι νομίζω θα μειωθεί ο αριθμός των δραματικών περιστατικών. Αλλά εγώ ευχαριστώ ε, να σας δώσω. Να, ευχαριστώ να δεχτώ και περισσότερες πληροφορίες αν έχετε. Και το γεγονό ότι αύριο θα έχουμε κάποια ε, πληροφόρηση για τα σχετικά ευρήματα νομίζω θα βοηθήσει και αν θέλετε επιπλέον ενημέρωση να κανονίσουμε μια συνάντηση για να δούμε και τα αποτελέσματα της αποστολής σας για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα Μετανάστευσης νομίζω πως ε, οτιδήποτε συνέβη μετά και τα όσα συμβαίνουν τώρα είναι επιβεβαίωση του γεγονότος ότι η ιδέα ότι έπρεπε να προτείνουμε ένα ολιστικό και συνολικό μοντέλο για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης εξακολουθεί να ισχύει. Και το έγγραφο αυτό που συντάχθη στην αρχή της θητείας αυτής της ε, Κομισιόν τη διακολουθούσε μία από τις δέκα κορυφαίες προτεραιότητες του Πρόεδρου Κιούνκερ για να παρουσιάσουμε ένα καλό έγγραφο. Το 2015 που είχαμε τα μεγαλύτερα νούμερα Καταλάβαμε ότι έπρεπε να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση των ικανοτήτων μας για να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες κρίσεις. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και μέχρι σήμερα. Οπότε, σίγουρα αυτή η μέρη σε διάταξη αποτελεί καθοριστικό στοιχείο. Και η ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου ακριβώς αυτό έδειξε. Και η επόμενη αυτό θα δείξει. Για πρώτη φορά λοιπόν τώρα έχουμε αυτήν ε, την επιχειρησιακή ικανότητα η οποία μπορεί να μην είναι απόλυτα βιώσιμη ήδη αλλά μπορεί να βοηθήσει τις χώρες εκείνες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κρίσης και που πρέπει να βοηθηθούν. Η Ελλάδα τώρα κάποια άλλη στιγμή θα είναι μια άλλη χώρα μέλος, οπότε ήδη αποτελεί αυτό μέρος αυτής ακριβώς της ημερήσιας διάταξης, αυτού του θεματολογίου. Και ανάλογα κάθε φορά θα κάνουμε. πήραμε όλοι μαθήματα από τα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αλλαγές πιο στοχευμένα και πιο γρήγορα για να βοηθούμε το σύστημα και την μεταναστευτική μας πολιτική έτσι ώστε να είναι πλήρης και να καλύπτει όλα τα στοιχεία και το θέμα των νόμιμων οδών μετανάστευσης, γιατί αυτή η νόμιμη μετανάστευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειωθεί η παράτυπη μετανάστευση. Ίσως όχι αυτή τη στιγμή που είμαστε σε κρίση, αλλά σίγουρα βραχυπρόθεσμα. Για το θέμα της επανεγκατέστασης, ε, resettlement, επειδή είπα ότι 81% είναι ήδη κάτι θετικό. Και πέραν αυτού, όλη η δουλειά που γίνεται τώρα στην νομοθετική διαδικασία για το σύστημα επανεγκατάστασης σαν κομμάτι του πακέτου για το άσυλο γίνεται προκειμένου να υποφαθούμε περισσότερο από τα μαθήματα που πήραμε μέχρι τώρα και από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Να μειώσουμε, ας πούμε, το διοικητικό άχθος και όλοι να μπορούμε να επωφελούμε από ένα καλύτερο σύστημα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στα πλαίσια αυτή τη νομοθετική δουλειά. Πάντω, η επανεγκατάσταση αυτή καθ' αυτή αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο σε σχέση με τι γενικότερε δεσμεύσει μα και το σύμφωνο για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες μετά τι συναντήσει Σούγκα που έγιναν πέρυσι. Θα δούμε τα αποτελέσματα του χρόνου. Και η επανεγκατάσταση αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων που αναλάβαμε κι εμείς. Στο νομοθετικό μας έργο εμπνεόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα για να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη να αποφύγουν και το διοικητικό άχθος στο θέμα της επανεγκατάστασης. Κοιτάω εδώ τις διάφορες σημειώσεις. Νομίζω ότι τα κάλυψα όλα. Α, ναι, στην αρχή είπα κάποια πράγματα για το καταπίστευμα. Πράγματι, για το Trust Fund, όντως υπάρχει θέμα οικονομικής στήριξης, αλλά πιστεύω ότι το όλο έργο του καταπιστεύματος και όλα τα προγράμματα και οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε θα έχουν αποτέλεσμα που θα εκτιμηθεί και θα αποτελέσει κινητήριο δύναμη για παρετέρω δράση. Έτσι καλλιώς στο ίδιο καράβι είμαστε όλοι. Οπότε με το κατεπίστευμα αυτό που θέλουμε να βοηθήσουμε την Αφρική, θα βοηθήσουμε και τους αυτούς μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κυρίες για τις ε, απαντήσεις σας και για την παρουσία σας πριν βεβαίως. Και σας, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε στις 9 ακριβώς με την διαχείριση της μετανάστευσης και για, την... και για τις επιστροφές. Ευχαριστώ πολύ.